Καλώ ήρθατε και πάλι αρχίζουμε τι εργασίε μα για το απόγευμα. Πρώτο σημείο, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η συγγήτριά μας για τι αλλαγέ ε, στην, ε, για τροποποίηση μάλλον του κανονισμού είναι η κυρία Στάουνερ. Σα ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κατά βάση χαιρετίζω τις προτάσεις Κομισιόν που μοίρασε με το πρόγραμμα ανάκαμψης ε, πριν από τα Χριστούγεννα για να καταπολεμηθεί η παγκόσμια οικονομική κρίση και είναι επίσης σωστό και αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα υπάρχοντα και να προσαρμοστούν σε αυτή την πρόκληση. Ήδη σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τις ανάλογες προσαρμογές που θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βεβαίως και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και να το προσαρμόσουμε κάπως. Θα δείτε πως έχω κάποιες τροπολογίες. Έχω βάλει και μια έκθεση, βεβαίω. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και συζήτηση με τον κύριο Σπίτλα, τον αρμόδιο επίτροπο χθες το βράδυ. Και για ακόμη μια φορά πιστήκαμε για τις προτάσεις της Κομισιόν και για τις δικές μου ιδέες Στόχος λοιπόν πρώτος πρέπει να είναι να γίνουν αυτές οι αλλαγές το συντομότερο δυνατόν γιατί όλα τα μέτρα βεβαίως δεν χρησιμεύουν σε τίποτα εάν δεν λαμβάνονται γρήγορα και νομίζω πρέπει πραγματικά να συμφωνήσουμε να καταλήξουμε στην πρώτη ανάγνωση σε ένα αποτέλεσμα αποδεκτό από όλους. Βεβαίως ξέρω ήδη από κάποιους συναδέλφους στην ε, ομάδα μου πως ε, έχουν κάπως διαφορετικές ε, ιδέες και αποκλίνουσες. Οπότε δηλώνω ευθύ εξ αρχή την ετοιμότητά μου να συζητήσω τα πάντα, όλες τις προτάσεις, όσο δυνατόν πιο γρήγορα και με ανοιχτό μυαλό. Όπως βλέπετε οι προθεσμία για τις τροπολογίες είναι ήδη την επόμενη Παρασκευή και όσοι θέλουν να υποβάλουν τροπολογίες να το κάνουν γρήγορα και ε, πριν ε, τελειώσει η προθεσμία ή δυνατόν. Υπάρχουν τέσσερα-πέντε σημεία εχμής στην αλλαγή του κανονισμού εδώ πέρα για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Γνωρίζετε πως εγώ προέρχομαι από μια χώρα που και στο Συμβούλιο από ό,τι μου λένε μαζί με άλλες χώρες που είναι έτσι καθαρής φορής έχει μια περιοριστική στάση όσον αφορά κάποιες αλλαγές αυτού του κανονισμού και αυτή η στάση για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων είναι και η δική μου στάση όσον αφορά βεβαίως το, το αποτελεσματικό κομμάτι. αυτό θα δείτε κάποιες ε, αλλαγές που έχω κάνει εδώ στην έκθεση. Αλλά, όπως σας είπα, μπορώ να, να συζητήσω τα πάντα. Θα αναφέρω μόνο κάποια σημεία επίμαχα το ύψος της χρηματοδότησης, του, το ποσοστό της χρηματοδότησης και της συγχρηματοδότησης πρέπει να μείνουμε στο 50% γιατί παρά ή μάλλον ακριβώς λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, καταστροφικής, υπάρχει ο κίνδυνος όταν παίρνει κανείς χρήματα ευρωπαϊκά να μην τα χρησιμοποιήσει πολύ αποτελεσματικά, απλά να τα χρησιμοποιήσει γιατί έρχονται και ρέουν. Μετά από κάποιες σκέψεις λοιπόν θεωρώ πως πρέπει να παραμείνουμε στο 50% ποσοστό της ε, κοινοτικής χρηματοδότησης και να μην πάμε ε, πιο πάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι συνάδελφοι βεβαίω από κάποια νοτιότερα κράτη έχουν διαφορετική άποψη όπως και οι σοσιαλιστές. Δεύτερον, οι αλλαγές αυτές ε, του κανονισμού θέλουμε να περιοριστούν όπως ε, προτείνει, πρότεινε και η Κομισιόν μέχρι τις 31 Δεκάτου 2010. Και αυτό το συζητάμε. Μία ουσιαστική αλλαγή του κανονισμού και το να πούμε ότι θα ισχύσει κάτι πέρα από την οικονομική κρίση είναι κάτι πρόημο αυτή τη στιγμή γιατί η εμπειρία από τα κράτη-μέλη με το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης δεν είναι τόσο μεγάλη. Τρίτον, πρέπει να πέσουμε κάτω από τον αριθμό των 500 όσον αφορά τις απολύσεις. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Να συμπεριληφθούν και οι, μικρο... και οι μικρές επιχειρήσεις και όχι μόνο οι μεγάλες βιομηχανίες. Και στο άρθρο 2 επίσης είναι και το ζήτημα σε ποιο χρονικό διάστημα έγιναν οι απολύσεις. Εκεί πέρα η Κομισιόν προτείνει 9 μήνες, εγώ ζήτησα 6, αλλά και αυτό το συζητάμε. Κατόπιν τα κατά αποκοπήν ε, ποσά είμαι θετική γιατί όπως κάναμε και στο κοινωνικό ταμείο πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και τα εμπόδια για να διατεθούν αυτά τα χρήματα το συντομότερο δυνατόν οπότε είμαι υπέρ της πρότασης της Κομισιόν δεν το βρίσκω τώρα για τα κατά αποκοπήν αυτά ποσά εν Νομίζω αυτά ήταν τα τα σημαντικότερα σημεία προς συζήτηση. Και εκεί πέρα υπάρχουν νομίζω και οι περισσότερες, θα υπάρχουν οι περισσότερες διαφωνίες, αλλά θα μείνω σε αυτά για να το συζητήσουμε και όλες περισσότερο. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Πολλοί θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Κοτινή, ο κύριος Σίλβα Πινέιντα. Κύριε Κοτινή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς ε, δηλώνω έκπληκτος ε, που υπέβαλε την πρόταση η Επιτροπή <laughs> για την τροποποίηση του κανονισμού. Ω επιτοπλίστων, πριν από δύο χρόνια η Επιτροπή μας, όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός, είχε υποβάλει μια πρόταση και στον ε, τριμερή άτυπο διάλογο απερίφθη η πρότασή μας από το Συμβούλιο. Ε, και μου κάνει εντύπωση που κατά τη διάρκεια τη τωρινή θητεία υποβάλλει αυτή την πρόταση η Επιτροπή. Υπό Βρετανική Προεδρίας 31 Δεκεμβρίου 2006 αποφασίστηκε ότι η χρηματοδότηση θα έχει ω ανώτατο όριο τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια. Και τελικά μείνανε ψίχουλα όμως. Ε, δεν φτάνουν ε, στους εργαζόμενους ό,τι μας περισσεύει εμάς ε. και 18 εκατομμύρια ευρώ μόνο καταναλώθηκαν, απορροφήθηκαν. Ναι. Ε, και γι' αυτό είχαμε κάνει και την πρόταση αυτή για να απορροβηθούν όντω αυτά τα κονδύλια. Τέλο πάντων, τα κριτήρια απονομή των κονδυλίων ε, είπε η Επιτροπή ότι δεν μπορούσαν να είναι λιγότερο αυστηρά και έπρεπε να απορροφηθούν τα κονδύλια. Είναι περίπλοκο ο μηχανισμό και είναι, παρά είναι αυστηρά τα κριτήρια. Ε, Χίλιου εργαζόμενου ε, ζητά η Επιτροπή, ενώ εμεί, η δικιά μα Επιτροπή, είχε ζητήσει 500 και στη διαπραγμάτευση προτείναμε 550, αλλά το απέριξε απέρριψε το Συμβούλιο και, εν πάση περιπτώσει, παρατηθήκαμε γιατί θέλαμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Επίσης ανάμεσα στις απολύσεις και στην παγκοσμιοποίηση, υπήρχε η σχέση βλέπουμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του Ταμείου και να απλουστεύσουμε την διαδικασία, να μειωθούν οι προθεσμίες. Ε, υπάρχουν διάφορα άλλα κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, αλλά σα λέω ότι το όριο είναι οι χίλιοι εργαζόμενοι και η βασικότερη μεταρρύθμιση έχει σχέση με το πρώτο που σα είπα, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη γραμμή του προπολογισμού για τη χρηματοδότηση, δηλαδή πρέπει να εγγράφεται στο κοινοτικό προπολογισμό και η χρήση θα είναι πολύ απλούστερη και δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να ασχολούμαστε και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Η αναθεώρηση πρέπει να βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, κατά παρέκκληση από τα βασικά κριτήρια παρέμβασης του Ταμείου, δηλαδή η σχέση με την παγκοσμιοποίηση, πέραν αυτό ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε στην ανακύκλωση όσων έχουν απολυθεί κατά παρέκκληση μέχρι το 2010. Συμφωνώ με αυτή την ιδέα και ε, το όριο πρέπει να κατέβει στους 500 εργαζόμενους από τους 1000 όπως ε, είπε η Επιτροπή επιτέλους αφού τους ή άλλους αυτό είχαμε προτείνει και εμείς και πρέπει να είναι πιο ελαστικοί κάποιοι κανόνες παραδείγματο χάρη να περάσουμε από 12 σε 24 μήνες για την εφαρμογή και ο χρηματοδότηση από 50% να πάει στο 75%. Συμφωνούμε απολύτως. Ε, και τα κράτη να συμμετέχουν μέχρι το 25% ούτω ώστε να εξετάσουν περισσότερου φακέλους. Γιατί ξέρουμε ότι ένα, όταν ένα κράτο δεν θέλει την παρέμβαση του ταμείου αυτού δεν υποβάλλει καν το φάκελο γιατί δεν έχει ε, κονδύλιο οπότε ε, δεν εξετάζουν καν πόσο εργαζόμενους έχει κτλ. Δηλαδή να, βάλουν, να συμμετέχουν σε μικρότερο βαθμό τα κράτη-μέλη για να εξετάσουμε περισσότερους φακέλους. Τώρα το θέμα των απολύσεων. Όταν εγκρίναμε αρχικά το έγγραφο είχε τεθεί το ζήτημα και η απόλυση δεν θα πρέπει να ε, περιορίζεται ε, στην ε, ειδοποίηση προς τον εργαζόμενο αλλά πριν την απόλυση αλλά και όταν η απόλυση είναι προϊόν διαπραγμάτευσης για, δηλαδή ε, όταν ε, παραδείγματος χάρη ανακοινώνεται για οικονομικούς λόγους ότι θα γίνουν απολύσεις. Ε, επίσης, ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, πάγια και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είχαν εκφράσει συνδυασμού για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, διότι δύσκολα μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μελλοντική τροποποίηση πρέπει να επιτρέψει την παρέκκληση, την παράταση μάλλον, για ένα επιπρόσθετο έτος όταν όμως προκύψει το θέμα και όταν θα είμαστε ε, σε, θέμα, σε θέση να, ε, να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Τροπολογίες 22 και 23 τώρα εφαρμογή σε κανονικές ε, περιπτώσεις δηλαδή η τακτική λειτουργία του Ταμείου και, εκεί ελοχεύει ένα κίνδυνο γιατί δεν θα δεχτούν τα κράτη-μέλη το περιεχόμενο αυτών των τροπολογιών. Αν θέλουμε συμφωνία για αυτές τις τροπολογίες πρέπει να αλλάξουμε στάση. Τώρα για τις των επιχειρήσεων χώρες με χαμηλότερου μισθού. Εντάξει, αυτό είναι ο λόγο που μεταφέρει τι δραστηριότητε τη μία επιχείρηση, αλλά όχι για άλλους λόγους. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό από το πεδίο εφαρμογής ε, του Ταμείου της παγκοσμιοποίηση, και ε, είναι και σχετικό το θέμα του χαμηλού μισθού. Ε, στην τροπολογία 11 προτείνω να περάσει η περίοδος ε, από 9 σε 6 μήνες ε, για, για την εφαρμογή του άρθρου 2β για κλάδους, όχι για μεμονωμένες επιχειρήσεις που καλύπτει το άρθρο 2α και συγκεκριμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ε από την εμπειρία βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται περισσότερο να δουν πόσες απολύσεις έχουν γίνει γιατί εμπλέκονται πάρα πολλές επιχειρήσεις μέσα σε ένα κλάδο. Τροπολογία 20, μείωση της περίοδου κατά την οποία θα πρέπει να υποβάλλεται ε, ε, η αίτηση από τη δημόσια διοίκηση από 10 έως ε, σε 8 εβδομάδες. Μα δεν είχαμε πρόβλημα με αυτό το, την περίοδο μέχρι στιγμής, οπότε δεν την υποστηρίζουμε. Τροπολογία 27, μείωση της περίοδου. Ε, εφαρμογής από 12 σε 9 μήνες ε, ε, θεωρούμε εμείς ε, αντίθετα ότι η πιο αποτελεσματική περίοδος θα είναι 24 μήνες. Πώς κάποιος που μειονεκτεί να βρει εύκολα θέση απασχόλησης και όσοι έχουν παραμείνει ένα χρόνο σε ανεργία δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο να βρουν θέση απασχόλησης. Ε, επίσης, μείωση της περιο... Ε, παράταση της περίοδου για την υποβολή αίτηση από την δημόσια διοίκηση και ε, για την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αυξηθεί σε 75%. Σα είπα και πριν πόσο σημαντικό είναι. Τόσο θα κλείσω, Πρόεδρε συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ταχθεί με το μέρος μας. Ωστόσο, ή άλλως ε, αυτό είχαμε ζητήσει εμείς ε, όταν είχαμε υποβάλει την ε, θέση μας στον τριμερή διάλογο από την ομάδα μας δεν θα υποβάλουμε τροπολογία και απευθύνω έκκληση να μην υποβάλουν ούτε οι συνάδελφοι για να καταλήξουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση και αυτό το, να προσαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστούμε κύριε Κοτινή. Ε, <laughs> Ξέρω πόσο σας καίει το θέμα. Όλους μας καίει αυτό το θέμα εξάλλου. Αλλά είναι τόσοι πολλοί που έχουν γραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε σύντομοι. Ξέρω ότι όλοι θέλετε να τοποθετηθείτε, αλλά παρακαλώ, έχουμε πάρα πολλού στον κατάλογο. 12-13 ομιλητέ έχουμε. Σίλβα Πινέντε και η κυρία Φιγκυρέιντο στην συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο δημιουργήθηκε μέσα σε κάποια συμφραζόμενα τότε θέλουμε να στηρίξουμε τους εργαζομένους που ε, ε, ε, πέφτουν θύματα μεταφοράς δραστηριοτήτων κάποιες επιχείρησης λόγω της παγκοσμιοποίησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντελήφθη ότι τώρα με την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει και με την προοπτική αύξηση της ανεργίας και την οικονομική κρίση θα πρέπει να τροποποιήσει το Παγκόσμιο Ταμείο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. και τα... καταλαβαίνουμε ότι θέλει να δώσει περιθώριο λιγμών μεγαλύτερη ελαστικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα εργαλεία που ήδη υπάρχουν, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με τις ε, ε τροπολογίες που υποβάλλει η κυρία Στάουνερ, παρότι τρέφω μεγάλο σεβασμό για αυτήν, διότι είναι πολύ περιοριστικές τροπολογίες ως προς τα ε, κονδύλια. Δεν μπορούμε με την τωρινή κατάσταση να ε, ε, είμαστε τόσο περιοριστικοί, δηλαδή θα πρέπει να ε, παρέχουμε κοινωνική στήριξη στους ε, απολυθέντες, έστω και αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές. Ε, επίσης είναι πήγον το θέμα, δηλαδή εντάξει εγκρίνουμε τις διατάξεις για το ΦΕΟΓΚΑ, για το Περιφερειακό Ταμείο, για το ΕΚΤΕ. Είναι πήγον το θέμα και να κινηθούμε και σε αυτό το τομέα και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Εγώ ε, προτείνω να την εγκρίνουμε ως έχει για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν έχω υποβάλει τροπολογίες και προτείνω και στους συναδέλφους ε, να μην υποβάλει κανένας τροπολογίες γιατί θα καθυστερήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πρέπει να ρυθμιστεί, να διεκπαιρεωθεί το θέμα το ταχύτερο δυνατόν. Αυτά ήθελα να πω εγώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Φιγκρέιντο και ο κύριος Πανσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σύντομη, πολύ πιο σύντομη από τον συνάδελφο Κοτίνι. Ε, δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ε, μέχρι στιγμής δεν έχει ε, εφαρμοστεί πλήρως, ε, δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως τα κονδύλια ε, του Ταμείου από τα 500 εκατομμύρια παραδείγματος χάρη που είχαν σχεδιαστεί αρχικά. Παραδείγματος χάρη το 2008 υπολείπονταν ακόμη 14 εκατομμύρια και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν πολύ αυστηρά, πολύ περιοριστικά και λυπούμεθα που ήδη τότε ε, δεν δέχτηκε η Επιτροπή να είναι ευρύτερο το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου και τώρα ε, ανακαλεί η Επιτροπή και η ίδια υποβάλλει αυτή την πρόταση για λόγους όπου είχαμε επικαλεστεί εμείς εκείνη την εποχή που είχε συγκροτηθεί το Ταμείο και είχαμε κάνει ε, σχετικές προτάσεις που είχε όμως απορρίψει η Επιτροπή. Θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία αν είχε δεχτεί τις προτάσεις μας η Επιτροπή. Συμφωνώ και με τον συνάδελφο, τον κύριο Σίλβα Πινέιντα, για την πρόταση της κυρίας Τάουνερ. Έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης ε, της κυρία Τάουνερ παρόλα αυτά και εάν εκείνη ε, μείνει στην πρότασή της ε, δεν μπορούμε παρά να υποβάλουμε προτάσεις ενίσχυσης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα σημεία που αναφέρατε εσείς συγκεκριμένα 24 ε, ε, μήνες ε, που εμείς είχαμε προτείνει 30, μέχρι στιγμής ήταν 30 μήνες. Η πρόταση της Επιτροπής για το 75%, εμείς θέλαμε 85% και τέλος πάντων κάποια άλλα σημεία όπου θεωρούμε ότι θα έπρεπε να την ενισχύσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Από την πορτογαλική εμπειρία επίσης μπορώ να σας πω για τις εδαφικές ζώνες Δηλαδή, ε, μία επιχείρηση ή περισσότερες επιχειρήσεις ε, του ίδιου κλάδου, του ίδιου βιομηχανικού τομέα να είναι στην ε, ίδια ζώνη, να είναι από την ίδια περιοχή. νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτεί η Επιτροπή γιατί το λέω. Στη Βόρεια Πορτογαλία υπάρχουν ε, παραδείγματος χάρη διάφορες περιοχές όπως της Μπέιρας. Έχουμε μικρές μισές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και δεν έχουν εναλλακτικέ λύσεις απασχόλησης οι εργαζόμενοι. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια διατύπωση χάρη στην οποία γρήγορα να ε, γίνουν ε, διαθέσιμα αυτά τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου της ε, Παγκοσμιοποίησης και θα κλείνοντας να πω ότι θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες που θα αναβαθμίσουν, θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πανσέρη και η κυρία Γιουκνέβιτς, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι κατανοώ ότι θα πρέπει ότι έχουμε, πορευόμαστε σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ιδιαίτερος ε, ανκαθόδης και είναι σημαντικό να φανούμε λίγο ευέλικτοι στις αποφάσεις μας. Και επίσης κατανοώ ότι πάντοτε είναι καλύτερο να έχουμε κάτι στα χέρια μας παρά απολύτως τίποτα στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αλλά ταυτόχρονα έχω την αίσθηση ότι η οικονομική κρίση ε, εξελίσσεται πολύ ταχύτερα από, ότι, από το ρυθμό που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και οι συλλαγές που κάναμε πριν από δύο χρόνια, για παράδειγμα, κατά κανέναν τρόπο δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα. Ούτε τα μέτρα που έχουν ληφθεί ανταποκρίνονται στην παρούσα κατάσταση. Νομίζω ότι οι αλλαγέ λοιπόν, οι μεταβολές που κάναμε δεν ε, επαρκούν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε τη δραματική κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά την αρχική πρόταση σε σχέση με αυτό το ταμείο, θα ήθελα να πω ότι παρουσιάσαμε επίσης κάποιες ε, τροποποίησεις και λάβαμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες βέβαια δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα δεν μπορούν παρά να είναι προσωρινές, έχουν έκτακτο χαρακτήρα και δυστυχώς αυτό δεν είναι λύση. Εγώ έχω μια κάπως διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι όλα αυτά δεν επαρκούν και θα ήταν χρήσιμο να κάναμε περαιτέρω αλλαγές. Ε, θεωρώ ιδιαίτερος ότι ε, θα πρέπει να αλλάξουμε το νόημα και τους σκοπούς αυτού του ταμείου. Νομίζω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ύψος των κονδυλίων και η Κομισιόν δεν έλεγξε καν γιατί δεν απορροφήθησαν αυτοί οι πόροι, αυτά τα κονδύλια. Νομίζω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να πάμε πέρα από αυτό που έχουμε ορίσει. Για παράδειγμα, στον αφορά τις απολύσεις. Δεν πρέπει να μόνο για συνοδευτικά μέτρα για τους απολυμένους, για τους απολυθέντες. Αλλά θα πρέπει να χράξουμε κάποιες πολιτικές, ώστε να μην φτάνουμε σε αυτές τις απολύσεις δεν είναι δυνατόν να περιοριζόμαστε στη συζήτηση συνοδευτικών μέτρων, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο πέραν τούτου να σχηματίσει κανείς μια ξεκάθαρη αντίληψη όσον αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και επίσης τα ενεργά συνοδευτικά μέτρα για την πολιτική της αγοράς εργασίας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εδώ μια συγκεκριμένη πεθαρχία όσον αφορά τις πολιτικές ομάδες, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επιβληθούν κάποιες τροπολογίες δεν είναι δυνατόν να το παρατείνουμε άλλο. Περιμέν... Δεν είναι εδώ να προβάλλουμε το επιχείρημα ότι αν υπάρχουν τροπολογίες θα καθυστερήσουμε. Νομίζω ότι είναι απολύτως χρήσιμο να υποβληθούν τροπολογίες και να γίνουν κάποιες αλλαγές. Η εναλλακτική λύση στην υποβολή τροπολογιών είναι είτε η Επιτροπή είτε οι πολιτικές ομάδες εδώ στην Επιτροπή και η δική μου πολιτική ομάδα να στηρίξει αυτή την απόφαση και στην περίπτωση αυτή αυτό θα αποβεί ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου και θα πρέπει εμείς να μεριμνήσουμε τα θέματα αυτά να συναδευτούν από μια απόφαση του Κοινοβουλίου. Η διεύρυνση αυτή να έχει συναδευτεί μια απόφαση του Κοινοβουλίου. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που επιθυμεί η Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν οι πολίτες τι γίνεται. Γιατί συνηθίζουμε να μιλάμε για μια κοινωνική Ευρώπη, αλλά όταν ε, ε, θέλουμε να την προωθήσουμε τελικά παραμένουμε στάσιμοι. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς αυτή η Ευρώπη δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή από τους πολίτες. Η κυρία και μετά ο κύριος Μάν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα κάποιες ε, συναντήσεις ε, με την Επιτροπή πρόσφατα και μιλήσαμε για τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, ότι είναι δηλαδή πολύ περιοριστικά και δεν δικαιολογούνται γιατί η πρώτη έκθεση έδειξε πως δεν γινόταν αρκετή χρήση του Ταμείου. Δεύτερον, γνωρίζουμε πως η αναθεώρηση αυτή, η πανεξέταση του Ταμείου έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι απολυμμένοι εργαζόμενοι χρειάζονται τη στήριξη, όχι μόνο λόγω της ε, παγκοσμιοποίησης, αλλά και λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο αυτή τη στιγμή πολύ επίκαιρο και αναβολή της συζήτησης αυτού του εγγράφου δεν ε, θα δικαιολογήσει την ύπαρξη αυτού του Ταμείου καθώς πρέπει να χρησιμοποιείται ακριβώς σε περιόδους κρίσεων όταν απολύεται ο κόσμος. Επίσης ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε στη μείωση του ποσοστού από το 75% στο 50% όπως προτείνει η κυρία Στάουνερ. Δεν είναι επειδή εκπροσωπώ μια χώρα που ε, θέλει αυτά τα λεφτά και την ε, συγχρηματοδότηση αλλά ε, είμαι υπέρ της υψηλότερης χρηματοδότησης από τα κοινοτικά ταμεία άρα δεν μπορώ να δεχτώ πλήρως αυτή την πρόταση γιατί τα χρήματα αυτά δείχνουν πως ε, το ταμείο αυτό είναι ένα από αυτά τα ταμεία που δείχνει αλληλεγγύη ε, και απτή με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάει πραγματικά τα λεφτά στον κόσμο. Σε σχέση με άλλα ταμεία, εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση, γιατί τα λεφτά αυτά πάνε μέσω ενδιαμέσων, αλλά τα λεφτά αυτού του ταμείου πηγαίνουν στο, στον κόσμο. Και αυτή είναι πραγματικά η ευρωπαϊκή ελληνική. Τώρα γιατί υποστηρίζω εγώ την περίοδο των 24 μηνών που προτείνει η Κομισιόν αντί για τους 10 μήνες που προτείνει η κυρία Στάουνερ. Το να βρει κανεί δουλειά σε 10 μήνες ε, με το τωρινό κλίμα την κατάσταση δεν είναι ρεαλιστικό. Το να επεκτείνουμε λοιπόν την περίοδο στους 24 μήνες είναι μια σωστή ε, και λογική απόφαση. Γιατί πρέπει ο κόσμος να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να βρει δουλειά και να λάβει στήριξη από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Είναι λοιπόν πραγματικά καλή αυτή η πρόταση. Μια πρόταση της εισηγήτριας που θα ήθελα να στηρίξω δεν έχει ίσως τόσο κέρια σημασία μάλλον θα συμφωνήσει η Κομισιόν είναι η τροπολογία 4 που θέλει η εισηγήτρια να διαγραφεί δεν νομίζω πως η Κομισιόν θα πρέπει να ζητήσει να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια για τεχνική αρρωγή ή άλλους ε, στόχους Οπότε η τροπολογία 4 είναι αρκετά καλή και η Κομισιόν δεν πρέπει να ζητάει περισσότερα λεφτά για τεχνική αρρωγή. Συνοψίζοντας, υποστηρίζω όλους τους κοιόδης εισηγητές που λένε πως η πρόταση της Κομισιόν είναι μια χαρά, δεν βλέπω εγώ κάποιο σοβαρό λόγο αναβολής της έγκρισης αυτού του εγγράφου. Πρέπει να βιαστούμε μάλιστα. Και άκουσα την πρόταση πως ε, πρέπει να χρηματοδοτηθεί ο ετήσιος προπολογισμός να είναι ένα δισεκατομμύριο. Αυτό θα είναι καλό για τους ευρωπαίους πολίτες. Ε, και αν το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει συνεισφέρει και στον καλυτερεύσουν οι ζωές τους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε ο κύριος Μαν και η κυρία Σρέντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα πράγμα πιστεύω ότι πέτυχε. Οι επιφυλάξει που είχαμε αρχικά όσον αφορά το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης ε, έγκυται στο ότι είναι μόνο μια προσπάθεια εξοραϊσμού. Το να πούμε δηλαδή στους εργαζόμενους ότι σας δίνουμε λίγα χρήματα στη διάθεσή σας και λύνει το θέμα. Νομίζω ότι όμως δοκιμάστηκε το πράγμα γιατί τα, πράγμα, τα κονδύλια αυτά αξιοποιήθηκαν και απέφεραν αποτελέσματα και νομίζω ότι σημειώσαμε τον τρόπο αυτό μια σημαντική επιτυχία και με τον τρόπο αυτό πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Είναι συγκεκριμένη μορφή ελεγγύης για τους, αυτούς που πλήττονται από αυτά τα προβλήματα και θέλουμε με περαιτέρω συνοδευτικά μέτρα, με μέτρα εκπαίδευση κλπ. να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αναπροσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ζαν ε, Λουκ, ε, πραγματικά μακρηγόρησε υπερβολικά. Αλλά νομίζω ότι ορισμένα σημεία τη έκθεση τη κυρία Φτάουνερ θα έπρεπε να τα υποστηρίξουμε. Ε, τον αριθμό 500 για παράδειγμα. αυτό θα πρέπει να το στηρίξουμε και θα πρέπει να μεριμνήσουμε να μειωθούν τα κονδύλια. Το 500 νομίζω ήταν σωστό. Έγιναν μακρές συζητήσεις σχέση με τις μικρές χώρες κλπ. Έχω ε, μια αλλαγή. τροπολογια 9 ότι αυτά είναι χρήματα για την ε, μεταεγκατάσταση, για την ε, μετατόπιση θέσεων εργασίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί η μετακίνηση αυτή να γίνει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέμε ότι πρέπει να περιεμφθεί το Ταμείο, γιατί πρόκειται για μια μείζωνα κρίση, τι θα γίνει για επιχειρήσεις όπου οι απολύσεις δικαιολογούνται σαν μια συνέπεια της κρίσης. Ε, δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια απάντηση. Γιατί είμαστε κάπως ασυνεπείς. Ε, δεν ξέρω, μέχρι στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις. Αν ε, η συζήτηση αυτή φτάνει, η σημερινή συζήτηση, για να πετύχουμε μια σύγκληση, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αυξήσουμε τα 500 εκατομμύρια σε ένα δις. Γιατί πρόκειται και ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν θα πρέπει οι χώρες μέλη να συγχρηματοδοτήσουν. Αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή υπεραξία και τα χρήματα αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι Ευρωπαίοι, Χωρί να χρειάζεται οι χώρε μέλη, οι άλλε χώρε να προσθέσουν κονδύλια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή βάση την οποία θα πρέπει να αποδεχτούμε. Ευχαριστούμε η κυρία Σουέντερ και μετά ο κύριος Ευχαριστώ. Το πρόβλημά μου είναι πως ε, ε, το ζήτημα εδώ πέρα είναι για ποια λεφτά μιλάμε. Δεν έχουμε καν λεφτά για αυτό το ταμείο. Είναι το αποθεματικό. Δηλαδή, εκεί όπου απομένουν σε κάποιο έτος χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γι' αυτό πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη για να είναι ξεκάθαρο. Και είχαμε συμφωνήσει τότε, είχαμε πει ναι. Εν τω μεταξύ βεβαίως προέκυψε το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν κάπου χρήματα γενικώ στον προπολογισμό, αλλά μιλάμε πάντα για χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή για τον χύψη λόγο δεν ξέρω, δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα του ΕΚΤ γιατί στην αρχή ήταν αργή η εκταμείευση μέχρι να ε, ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κτλ. Υπήρχαν κονδύλια διαθέσιμα και από όσο ξέρει η Κομισιόν μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έπαιρνε μέχρι στιγμή λεφτά. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση όπου δεν παίρναν λεφτά ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ταμείο ή από το Ταμείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, αλλά από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και επίσης για το σχέδιο ανάκαμψης, αλλά αυτή η κατάσταση δεν θα ισχύει στο μέλλον, γιατί πρώτα απ' όλα ε, πηγαίνουν ε, στον τομέα της ε, άφρυνσης, στον διευκολύνσεων και από την άλλη μεριά το να προσπαθήσουν, προσπαθούν δύο κανονισμοί να πάρουν λεφτά από το ίδιο ταμείο, πρόβλημα που δεν έχει ακόμα λυθεί. Έτσι ώστε για να έχει, πρέπει να έχει και κάποιο νόημα η κατάσταση και να μην έχουμε και ανταγωνισμούς ε, επιτόπου, εκεί όπου θα εκταμιευτούν τα λεφτά, δηλαδή άνθρωποι στην κατάσταση που περιέγραψε ο κ. Πασέρη και ή να ανταγωνίζονται ξέρω εγώ με τους μακροχρόνια ανέργους για το ποιο δικαιούται τα λεφτά αυτά επειδή είναι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οπότε όταν μιλάμε για αύξηση ε, του ποσού, μιλάμε για αύξηση ενός φανταστικού ποσού που δεν προβλέπεται κάπου στον, στον προϋπολογισμό. Πολύ απλά δηλαδή, de facto λέμε ότι το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης θα πάρει περισσότερα λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό σημαίνουν αυτά που λέμε, να το ξέρετε. Οπότε, εγώ θα ήμουν πολύ ε, προσεκτική και το ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα λεφτά ούτε αυτό ισχύει. Στα διαρθρωτικά ταμεία υπάρχουν αυτά τα λεφτά μέχρι το 2013. Έχουμε ακόμα καιρό. Δηλαδή αυτό το οποίο εικονικά κάθε χρόνο παίρνουμε από το απόθεμα θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αν είχαν εργαστεί αναλόγως και τα κράτη-μέλη. Να το ξέρουμε αυτό. Δεύτερον, που για μένα είναι εξίσου επικίνδυνο και που η Κομισιόν εδώ πέρα λίγο το το σκέπασε και δεν έλαβε υπόψη ε, αυτά τα οποία είπε το Κοινοβούλιο αφορά τη μετατόπιση επιχειρήσεων εντός όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι αποτελέσματα έχει αυτή η μετακίνηση. Η μετακίνηση και θα ήθελα μία απάντηση για το πώς σκοπεύει η Κομισιό να εμποδίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μία επιχείρηση να πηγαίνει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και να προσπαθεί να έχει αυτά τα θετικά αποτελέσματα της μετακίνησης. Γιατί εμείς θέλουμε να υποφεληθούν οι εργαζόμενοι από αυτά τα, τα χρήματα. Και επίσης τα κοινωνικά σχέδια που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις και αποτελούν μέρος των διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους πώς θα τηρηθούν από τις ε, επιχειρήσεις για να έχει ένα επιπρόσθετο αποτέλεσμα αυτό το δημόσιο ταμείο που είναι και ο στόχος τελικά. Γι' αυτό νομίζω πως ε, προς τα εκεί στοχεύουν και οι τροπολογίες μου. Εγώ ανήκω σε αυτούς όπως κυρία Στάνερ και ο πρώτος που ασχολούμαστε συνεχώς με αυτά τα πράγματα και βλέπουμε διάφορα πράγματα κατά καιρούς τα οποία περνάει η Κομισιόν, δηλαδή έχουν κατατεθεί εδώ πέρα τροπολογίες που πηγαίνουν πέρα από τον τωρινό κανονισμό και παρόλα αυτά περνάνε όπου παραδείγματος χάρη είναι εις βάρος ε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων τα κονδύλια τα οποία εξασφαλίζονται και εδώ πέρα δεν έχουμε πολύ καλές διατυπώσεις δηλαδή πάντα λέμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εδώ ένα συνδυασμένος ε, μισθός και να μην υπάρχει μια επιδότηση αν θέλετε ε, των μισθών. Απλά να ε, συνεχίσουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια εκπαίδευση κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Είναι προβλήματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε να μην συμβούν. Γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε τις διατυπώσεις εδώ και Εξού και η τροπολογία για την τεχνική αρρωγή της κυρίας Γιουχνεβιτσένε που την υποστηρίζουμε είναι πολύ σημαντική. Αυτό το οποίο είπε επίσης η κυρία Στάνορ ότι έχουμε μια υποκατάσταση ξαφνικά της δημόσιας διοίκησης. Και θα είχε περάσει κάτι τέτοιο εάν δεν υπήρχαν βεβαίως οι έντονες ε, διαμαρτυρίες μου. Οπότε Πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά πολύ λεπτομερώς και δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θέμε τώρα εμείς τροπολογίες στην πρόταση Κομισιόν. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και σημαντικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για το πού πηγαίνουν τα χρήματα, αν πηγαίνουν εκεί που θέλουμε εμείς να πάνε, αν θα πάνε σίγουρα, αν διατηρείται η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αν έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα ζητήματα και μόνο υπ' αυτές τις ε, ε, προϋποθέσεις και γι' αυτό το λόγο άλλωστε καταθέτω αυτές τις ε, τροπολογίες. Νομίζω υπάρχουν και τροπολογίες της κυρίας Στάουνερ γιατί και εκείνη ασχολείται συνέχεια με αυτά τα ζητήματα που έρχονται από τα, τα κράτη-μέλη. Και δεν ξέρω πραγματικά εάν όλα αυτά έχουν πάει στο σημείο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποβί, ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι λίγο σουρεάλ η κατάσταση. Αναθεωρούμε τον κανονισμό για ένα ταμείο που δεν λειτουργήσε. 3% απορρόφηση κονδυλίων μόνο. Επειδή υπάρχει κρίση, έτσι λένε. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, δεν πρέπει να καταλάβουμε πρώτα γιατί δεν λειτουργήσε ο κανονισμός. Δηλαδή ποσοτικά από πλευράς απορρόφησης σαφώς αποτύχαμε. Και το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, Ούτε και ποιοτικά δεν ξέρουμε αν ήταν ε, επιτυχέ το εγχείρημα. 18 εκατομμύρια ευρώ απορροφήθηκαν, λέμε. Ωραία, πού πήγαν Ήδη αυτά τα δύο χρόνια που λειτουργεί το Ταμείο πήγαν τα λεφτά στους ενδιαφερομένους εργαζόμενους. Εγώ θα ήθελα μια απάντηση γι' αυτό. Να υπενθυμίσω, Πρόεδρε, και στους συναδέλφους αυτά που έλεγα στις 12 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια. Περιμένουμε ένα σύστημα με παραγωγική δράση για επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, λαμβάνοντα υπόψη τα αποτελέσματα του φόρουμ για, για τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Είναι σουρεαλιστική η συζήτηση, Πρόεδρε. Λέμε θα, ψηφίσουμε, θα υπερψηφίσουμε ή θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες για περισσότερα χρήματα, περισσότερο χρόνο κτλ. Υιοθετώντα το, είτε το σύστημα της Επιτροπής είτε το σύστημα της κυρίας Τάουνερ με τις τροπολογίες, αλλά, συγγνώμη, οι δικοί μας οι στόχοι των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπληρώνονται. Ε, δεν είμαι καθόλου πεπισμένος. Θέλουμε να παρεμποδίσουμε τη διαδικασία ή θέλουμε να την προάγουμε. Το είναι ένα ε, βασικό ερώτημα. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως θέλουμε να συνεχιστεί η διαδικασία. Ε, λοιπόν, ασυζόμενος αυτό θα κάνω δύο προτάσεις. Ε, πρώτον, για να ληφθεί υπόψη η γενικότερη κατάσταση, ας μην υποβάλουμε τροπολογίες, ε, ας ακολουθήσουμε τη γραμμή της Επιτροπής. Όπως είπε ο Ζαν και άλλοι, γιατί και εγώ ήμουν σκιώδης, με τον συνάδελφο συνεργάστηκα πριν από δύο χρόνια για αυτό το θέμα. Η Επιτροπή μας λέει τα ίδια που προτείναμε εμείς πριν από δύο χρόνια. Θα, συγγνώμη, αλλά θα ήταν... Θα ήμασταν ε, αχάριστοι να μην ε, τα δεχόμασταν. Έχω δύο προτάσεις που τις είπε και ο κύριος Πανζανή. Ένα λεπτάκι. Πρόταση ψηφίσματος πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μια ενεργό πολιτική απασχόλησης άσχετα αν δίνουμε εκατομμύρια, 500 ε, εκατομμύρια ή ένα δις, 10 ή 12 μήνες, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι επιθυμούμε μια ενεργό πολιτική απασχόλησης, να μην παρεμποδίσουμε τη διαδικασία. Και άρα δεν χρειάζονται τροπολογίες, ψήφισμα χρειάζεται, δεύτερη υποπρόταση ας την πω έτσι. Να έχουμε συμφωνήσει και με τον Λουί. Τριμερή άτυπο διάλογο πώς θα οργανώσουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ούτω ώστε το θέμα της ποιότητας να ληφθεί δεόντως υπόψη. Λοιπόν, α μην κολλησιεργούμε. Α εγκρίνουμε τις προτάσεις της Επιτροπής, ένα πρώτο αυτό και δεύτερον, ας εκφράσουμε τις απόψεις μας μέσα από ένα ψήφισμα και μέσα από ένα τριμερή άτυπο ε, διάλογο. Ο κύριος Χάσε Φερέιρα και μετά ο κύριος Στέφεν Χιούς. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δύο είναι τα βασικά ζητήματα κατά με σε αυτό το στάδιο. Με την ιδιότητα του βουλευτή και με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη ενδιαφέρομαι για αυτά τα δύο ζητήματα. Πρώτον, Ε, υπάρχουν διάφορα παραδείγματα εφαρμογής. Εγώ ένα που γνωρίζω ε, δείχνει ότι ήταν πολύ χρήσιμο το Ταμείο και οι εργαζόμενοι δεν είχαν ε, καθόλου ενδιασμού επιφυλάξει σχέση με την εφαρμογή του Ταμείου, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν, παροφήθηκαν σωστά τα κονδύλια. Ε, από τι πληροφορίε που έχω, πήγα εγώ επί τόπου, είδα τα εργοστάσια που κλείσανε και ε, η Γκαμπριέλα Στάουνερ με την ευφυΐα και την ευελιξία που την χαρακτηρίζει σίγουρα έχει υποβάλει πολύ καλές τροπολογίες και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι σε σχέση με την τροποποίηση του κανονισμού. Τώρα, εάν υπάρχει ε, διαθεσιμότητα των κονδυλίων, λέμε ότι θα περάσουμε από 50% σε 75% αλλά το 75% είναι το ανώτατο όριο. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει ότι υπολείπονται κονδύλια. Δηλαδή είναι θέμα ότι μπορούμε να ξοδέψουμε μέχρι το 75%. Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε όχι να προτείνουμε 80-85%. Μα όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει το 75% και ε, δίκιο έχει εγώ που συνήθως απευθύνω επικρίσεις για αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι λογικό λογική ε, η πρόταση της Επιτροπής. Ε, εφόσον ανεβαίνει το ποσοστό από το 50% πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική μας κατάσταση για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ε, και ε, συμφωνώ λοιπόν με τους συναδέλφους και τους κατανοώ γιατί πρέπει να ικανοποιήσουν και τους ψηφοφόρους του. Αλλά ε, μην ξεχνάτε ότι θα επιδεινωθούν ε, τα προβλήματα ε, λόγω της ανευθυνότητας στην δημοσιοοικονομική διαχείριση στη ΣΥΠΑ και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όπως λέει με σύνεση η Επιτροπή, θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό το ποσοστό της συγχρηματοδότησης. Για την προθεσμία τώρα, σε κάποια κράτη-μέλη ανταλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάουσες καταστάσεις, ε, ότι σε κάποια κράτη-μέλη έχει ήδη εφαρμοστεί η διαδικασία και έχουν εμπειρία. Ε, σε κάποια άλλα δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και άρα θεωρούν ότι θα είναι περίπλοκη η διαδικασία. Θυμηθείτε τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής και παρέμβασης του Ταμείου και προτείνεται η μείωση της προθεσμίας αλλά τέλος πάντων εάν θέλετε αν κρίνουμε από την εμπειρία ε, ήταν πολύ καλή η χρήση του Ταμείου και θα επιδεινωθεί η κρίση. Συμφωνώ και με τις ανησυχίες του Πιέν Αντώνιο Πανσέρη μπορούμε να εγκρίνουμε αυτό ένα ψήφισμα ε, για την ενεργοπολιτική απασχόληση. Αλλά ας μην παρεμποδίσουμε τη διαδικασία, συνάδελφοι, γιατί σε λίγους μήνες θα σταματήσει να λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Θα ε, γίνουν ριζικές αλλαγές εδώ. Ε, υπάρχουν πράγματα ε, που κάναμε το 2007, το 2008 που δεν μπορέσουμε να κάνουμε το 2010. Ε, εγώ λέω να διατηρήσουμε το 75% που προτείνει η Επιτροπή, να διατηρήσουμε τον αριθμό των μηνών που προτείνει η Επιτροπή και εντάξει για τα προβλήματα εφαρμογής ας ε, ε, εξυγχρονίσουμε τη διαδικασία, ας κατονομάσουμε τα προβλήματα, αλλά ας μην παρεμποδίσουμε τη διαδικασία από πλευράς μας. Ε, δεν πρέπει το Κοινοβούλιο να απόσχει από την στήριξη αυτής της διαδικασίας που δεν σχετίζεται μόνο με την παγκοσμιοποίηση αλλά την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης λόγω της ανευθυνότητας στους χρηματοπιστωτικούς κύκλους τον είπα, και της Ευρώπης. Ε, και ε, σχετικά με το ψήφισμα σίγουρα θα ήταν πολλοί που θα υποστήριζαν αυτή την ιδέα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που έχουν πέσει θύματα αυτής της κρίσης και δεν φέρουν καμία ευθύνη, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ξεκρέμαστους. Ευχαριστούμε ο κύριος Στίφεν Χιούς ε, και η κυρία Λίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω τα όσα ακούστηκαν. Συμφωνώ με όσους είπαν πως δεν πρέπει να καθυστερήσουμε αυτή την πρόταση. Θα θυμάστε τι έγινε και στην συνεδρία των συντονιστών. Εγώ είχα πει πως πρέπει να το δούμε χωρίς τροπολογίες όπως πρέπει και οι κανηγιώνες για το ε, κοινωνικό ταμείο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Οπότε απογοητεύτηκα που άκουσα πολλούς, ε, πολλές τροπολογίες πολύ περιοριστικές της εισηγήτριας. Ελπίζω να το ξανασκεφτεί και να σκεφτεί έστω και αυτή τη στιγμή να τις αποσύρει κάποιες αν όχι όλες. Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να το εγκρίνουμε αυτό γιατί η κρίση είναι τώρα συμβαίνει και πρέπει να προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Νομίζω η ιδέα του κυρίου Παντζήρη και του κυρίου Μποκίλε, Να περάσει η πρόταση και μετά να δούμε τη δυνατότητα ψηφίσματος εάν είναι δυνατό κάτι τέτοιο για να, περάσει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ε, ίσως αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Ευχαριστούμε η κυρία Λίν και ο κύριος Δησιέμ. Ναι, ευχαριστώ. Θα είναι σύντομη. Και τίνω να συμφωνώ με τον Στίβεν ότι με τις ε, τροπολογίες που κατέθεσαν από την εισηγήτρια, ιδιαίτερα στην 11, 26 και 27, ε, συμφωνώ. Α, δεν κατάλαβα γιατί στην 11 αλλάζει η περίοδος ε, από 11 μήνες σε 7 μήνες όσον αφορά τις απολύσεις. Επίσης η αύξηση του 50% στο 55% δεν έχει νόημα. Βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση και θέλουμε να έχουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε, το ταχύτερο δυνατό, να φτάσουν τα χρήματα αυτά στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Τώρα για την 27. Δε, 10 μήνες από 24 μήνες που προτείνει η Επιτροπή και πάλι δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό που κρύβεται από πίσω. Θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα όσο απλά γίνεται και όσο πιο εύκολα να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά και όπου τα χρειάζονται. Αν δεν μπορέσετε να αποσύρετε ορισμένε από τι τροπολογίε σα, θεωρώ ότι οι υπόλοιποι από εμά δεν θα αισθανθούν, την... θα αισθανθούν στην ανάγκη να υποβάλουν τροπολογίε, Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουν όλε οι πολιτικέ ομάδε να συμφωνήσουν επί μια ενιαία στρατηγικής. Ευχαριστούμε κύριο Ντισί. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω, όπω ε, πολλοί άλλοι συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστέ, ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να εισβάλλει με το πιο χρήσιμο τρόπο, να εισφέρει με το πιο χρήσιμο τρόπο σε μια κατάσταση όπου πολλοί εργαζόμενοι σε βιομηχανίε αντιμετωπίζουν όχι μόνο αναδιαρθρώσει που υπήρχαν άλλωστε και πριν από την κρίση και συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι αντιμέτωπη μια κρίση τη ίδια τη παγκοσμιοποίηση που πλήττει την αυτοκινητοβιομηχανία ιδιωτέρω αλλά και πολλού άλλου κλάδου. Οι αρχέ είναι σωστέ. Ε, και αν ε, πολλοί από εμά θεωρούσαν στην αρχή ότι τα κριτήρια ήταν ιδιαίτερα περιοριστικά, πιο περιοριστικά από ό,τι θέλαμε. Και η υλοποίησή τους ήταν απογοητευτική, γιατί τα ποστά απορρόφησης το αποδεικνύουν οι ορισμένε απόψει η πρόταση τη Κομισιόν σήμερα ε, υιοθετεί τι αρχικέ προτάσει τη δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή. Προφανώς ορισμένα μέλη θα ήθελα να πάει πιο πέρα η Κομισιόν και κατανοώ πολύ καλά την αντίδραση του κ. Πανσάρη. Ε, μπορεί κανεί να διαρωτηθεί εάν δεν θα έπρεπε ίσω να ξανασυζητήσουμε το κοινωνικό ε, θέμα εδώ. Πρόκειται για ένα, γιατί πρόκειται για ένα ταμείο κοινωνική υποστήριξη όσον αφορά τι συνέπειε τη κρίση και τη χάραξη μιας ενεργού πολιτικής απασχόλησης που να μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο το φαινόμενο της παγκοσμιοποίηση, αλλά και τι συνεχεί εξελίξει στον χώρο της βιομηχανίας και ιδιαίτερα όσον αφορά αυτή την κατεπίγουσα ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση. Κύριε Παζάρη, ανοίξτε τον δρόμο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε μια ψήφ, ένα ψήφισμα που θα μας επέτρεπε να ανοίξουμε πάλι με την Επιτροπή μια εισβάθος συζήτηση για τις εξελίξεις και άμεσα χωρίς να χάνουμε χρόνο με τροπολογίες που είναι λίγο επίμαχες να υιοθετήσουμε το όραμα του κανονισμού Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια παρατήρηση. Εάν δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που ενελοποιούν ε, στέρεους μηχανισμούς υποστήριξης, είναι προφανές ότι οι χώρες μέλη θα μπουν στον πειρασμό να κινητοποιήσουν τα δικά τους υποστηρικτικά μέτρα. Βλέπουμε τι γίνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία και θα ανακύψουν στην περίπτωση αυτή προβλήματα διαστρέβλωσης του ανταγωνισμού έστω και αν πρόκειται για κοινωνική υποστήριξη. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε ένα μεγαλύτερο τμήμα του Ταμείου να μπορεί να κινητοποιηθεί με κριτήρια πιο ευέλικτα. Έστω και αν εκ παραλίλου ε, ξεκινήσουμε μία συζήτηση εις βάθος. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πω και εγώ δύο πράγματα. Όπως είπε ο κύριος Χιούς, το συζητήσαμε και με τους συντονιστές το θέμα στη Σουηδία. Λέμε σε μία παροιμία ότι όσο εμείς συζητάμε ε, ένα πρόβλημα, αυτό αυξάνεται. Έχουμε πρόβλημα αυτό το πρόβλημα η πολιτική, ότι δηλαδή έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση που περιέγραψε πολύ σωστά ε, ο κύριος Πινέιντα ε, και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν θα μας καταλάβει κανείς που ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Ε, δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε πιο γενναιόδοροι ή πιο περιοριστικοί. Υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων και μπορούμε να συζητάμε. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά ας το ζυγίσουμε αυτό ε, και ας ε, σε σχέση με αυτά που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη που βρίσκονται σε μια δυσχερή κατάσταση. Και υπάρχει το θέμα του, του του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, και ήταν πολύ καλή απόφαση που πήραμε, που δεν υποβάλαμε τελικά τροπολογίες. Θα μπορούσαμε και να το είχαμε κάνει, αλλά τα ζυγίσαμε καλά τα πράγματα και αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τώρα το ίδιο ζήτημα τίθεται και με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης άσχετα με ποιο ταμείο είναι, το κοινωνικό ή το ταμείο προσαρμογής. Τέλος πάντων είναι μικρά εργαλεία ακόμη και αν υποβάλουμε τις τροπολογίες. Δεν είναι αυτό το σημαντικό για ποιο ταμείο μιλάμε. Το σημαντικό είναι να περάσουμε εμείς οι πολιτικοί ε, αυτό το σημαντικό μήνυμα στα κράτη μέλη ότι και εκείνα πρέπει να δράσουν γιατί φέρνουν την πρώτη στη ευθύνη στη, στα πλαίσια της κρίσης. Εμείς τι εργαλεία έχουμε. Έχουμε το κοινωνικό ταμείο και έχουμε και το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Είναι περιορισμένα μεν, σημαντικά δε για τους πληγέντες. Ε, και είναι σημαντικά γιατί περνάνε το μήνυμα αυτό που σας είπα στα κράτη-μέλη, που να δράσουν και εκείνοι. Κίνα. Εντάξει, συμφωνώ ότι μπορούμε να συζητήσουμε διεξοδικότερα το θέμα, αλλά να κολυσιεργήσουμε. Αξίζει αυτό γιατί θα περάσει η ευκαιρία. Έχει ήδη, υπάρχει ήδη η κρίση, έχουν απολυθεί οι εργαζόμενοι. Μας απευθύνουν επικρίσεις διότι δεν ε, αντιδρούμε. ας μην μας κατηγορήσουν ότι καθόμαστε και συζητάμε τώρα πόσους μήνες θα κρατήσει και τι ποσοστό θα έχουμε ε, αντί να κάνουμε κάτι στην πράξη. Ακούστηκε η πρόταση ότι καλύτερα είναι να εκδώσουμε ψήφισμα. Μπορεί. Ε, το πρωί που στη ψηφοφορία για τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση ε, είπαμε ότι ε, υπό το φως της σοβαρότητας της οικονομικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να λάβει έκτακτα μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της ε, ευρύτερης ε, πρόσβασης στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να επικουρήσει τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε διάφορες δύσκολες ε, καταστάσεις όπως αυτοί που είχαν προσωρινή θέση αποσχόληση και έχουν απολυθεί και τα και τα υπερψηφίσαμε αυτά το πρωί. Αυτά κάναμε στην ψηφοφορία για τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης, οπότε είναι αναμενόμενο να ακολουθήσει αυτό το δρόμο η Επιτροπή. Δεν μπορεί το άλλα να λέμε το πρωί και άλλα το απόγευμα. Το ίδιο μήνυμα θα πρέπει να περάσουμε. Και ελπίζω θα ανταποκριθεί η Επιτροπή σε αυτά που εμείς αποφασίσαμε και εγκρίναμε το πρωί. Επιτροπή. Η uh, e πρόταση της ε, Επιτροπής για... Ε, είναι τμήμα της, ε, του προγράμματος ανάκαμψης το οποίο παρουσιάστηκε πέρσι και το οποίο υιοθετεί μια σειρά μέτρων τα οποία είναι ακριβή, περιορισμένα στο χρόνο και στοχευμένα σε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτή η πρόταση ευθυγραμμίζεται πλήρως με την προσέγγιση αυτή. Και για το λόγο αυτό η Επιτροπή εξέφρασε την επιθυμία να δει, ε, να εγκρίνονται ταχαίως αυτές οι τροπολογίες, ούτως ώστε σύντομα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το εργαλείο σε σχέση με την κρίση. Ε, κάναμε μία σειρά επιλογών σε σχέση με το τι θα πρέπει να αλλάξει και ε, ποια θα είναι η δυνατότητα διεύρυνσης των δυνατοτήτων που έχουμε και πραγματικά ήρθαμε, όπως είπαμε, μια πρόταση που είναι στοχευμένη και περιορισμένη στο χρόνο. Ε, το κάναμε αυτό μετά από συζητήσεις με τις χώρες μέλη. Ζητήσαμε, ρωτήσαμε τις χώρες μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους πού βρίσκονται οι δυσκολίες, πού βρίσκονται τα όρια, πού βρίσκονται τα εμπόδια στην χρησιμοποίηση των κονδυλίων, στην απορρόφηση των κονδυλίων. Τους ακούσαμε και καταλήξαμε ε, συμπεριλαμβάνοντας τις ιδέες αυτές που παρουσιάστηκαν και από τις χώρες μέλη και από τους κοινωνικούς εταίρους. Επίσης εξασφαλίσαμε το Ταμείο να συμπλέει ή να ευθυγραμμίζεται μάλλον με την αρχική ιδέα του Ταμείου, δηλαδή να υποστηρίζει τους εργαζόμενους που απολύθησαν στην επία της παγκοσμιοποίησης. Παραμείναμε σε αυτό το όριο, δηλαδή θέλησαμε να διαθέσουμε χρήματα για τους απολυθέντες. Ελπίζω ότι οι προτάσεις αυτές πραγματικά θα διευκολύνουν αυτό το έργο και ε, σας τις υποβάλλω λοιπόν να τις εξετάσετε. Ευχαριστούμε. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Στάουνερ για να λήξει και η συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις. Ε, αυτά τα οποία είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα. Σύντομα θα αναφερθώ σε κάποια πραγματάκια. Συνάδελφος Φιγερέδο έφυγε. Πρέπει να ξεκαθαρίσω πως ε, αυτό το οποίο λέει και η Κομισιόν, δηλαδή μέχρι στιγμής δεν είχαμε περιοριστική χρήση του Ταμείου. Ήταν και εδώ πέρα η συνάλφος ε, Σερεντερίδα με κάθε τροπολογία και θα σας το πω ξεκάθαρα, πάρα πολύ το είδαν αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε, τα μικρά αυτά ποσά τα οποία εκταμιεύτηκαν τα 18 εκατομμύρια δεν οφείλονται σε κάποια περιοριστική τακτική. Τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Είναι άλλα ζητήματα τελευταία που δεν θέλω να τα αναφέρω. Πρόκειται απλά για ένα νέο μέσο. Πρέπει να το αντιληφθούν και τα κρατημέλη και να το εφαρμόσουν και παίρνει αυτό λίγο χρόνο. Οπότε η Κομισιόν μπορεί να τα επιβεβαιώσει αυτά. Ζητήσαμε πράγματα όπως οικογενειακά επιδόματα που απομακρύνονται πολύ από το σκοπό του Ταμείου και δεν θα θέλαμε και στο μέλλον να τα κάνουμε γιατί με αυτό το μέσο δεν πρέπει να απαλλάξουμε τα κράτη-μέλη από τις υποχρεώσεις τους για να δίνουν κοινωνικές φορές και για οικογενειακά επιδόματα δεν είναι αυτός ο ρόλος μας εδώ πέρα. Τώρα συμφωνώ με τον συνάδελφο Παντσέρη πλήρως πως ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης δεν φτάνει για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Είναι πράγματι σταγόνα στον ωκεανό και δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες ε, προσδοκίες ή να δημιουργήσουμε τέτοιες προσδοκίες. Αυτό το οποίο θα χρειαζόμασταν, συμφωνώ πλήρω, το είπε πολύ ωραία, χρειαζόμαστε μια πολιτική ή πολιτικές έτσι ώστε να μην καταλήγουμε καν σε τέτοιες μαζικές απολύσεις, αλλά έτσι, από αυτό απέχουμε και σε αυτό το κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη απέχουν γιατί η κοινωνική διάσταση αυτής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης δεν ε, υπάρχει, δεν ε, λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε. Το λέω αυτό πάντα βεβαίως ε, προς την Κομισιόν που πάντα με τις επιχειρήσεις ασχολείται και ελάχιστα με τις ανάγκες των εργαζομένων. Ποιο ήταν το επόμενο, ναι. Ε, η μείωση από τους 24 στους 10 μήνες. Κοιτάξτε, με αυτό το ταμείο κατά της παγκοσμιοποίησης, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είχαμε ποτέ την πρόθεση να έχουμε μια διαρκή επιδότηση. Μιλάμε για μια βραχυπρόθεσμη παρέμβαση κρίσης. Δεν θα προωθήσουμε εδώ πέρα τους μακροπρόθεσμα ανέργους. Δεν ξέρω τι γίνεται στις δικές σας χώρες και πώς ορίζονται οι μακροχρόνια άνεργοι, αλλά για μένα 24 μήνες είναι μακροχρόνια άνεργοι και αυτοί υποστηρίζονται και καλά μάλιστα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εκεί υπάρχουν τα μέσα και στο πλαίσιο αυτό ακριβώς τίθεται ζήτημα συμβατότητας με το κοινωνικό ταμείο, το είπα και πριν. Δεν θέλω εγώ αυτά τα δύο μέσα να μπλεχτούν και τελικά κανείς να μην ξέρει τι πρέπει να, να χρησιμοποιήσουμε ή μήπως υπάρχει κάποια διπλή ενίσχυση. Ο Τόμας Μαν έθεσε το ζήτημα του ορισμού το οποίο το όρισε ως παγκοσμιοποίηση. Ε, υπήρχε αυτό και στο παρελθόν. Γιατί η παγκοσμιοποίηση είναι τα πάντα. Δηλαδή ο καθένας καταλαβαίνει και ό,τι θέλει με την ε, παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχει και κάποιος ορισμός. Δεν ξέρω, α, τα κατεβαίνει η οθόνη, θα δείξετε εδώ τον ορισμό της παγκοσμιοποίησης. Καλό θα ήταν. Ε, αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα και εντάξει αναμένω προτάσεις από όλους σας γι' αυτό πράγματι. Η συνάδελφος Σρέντερ είπε πως είναι και το ζήτημα της μετατόπισης των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης και να ζητάνε τα ίδια κονδύλια. Όλοι γνωρίζουμε πως ε, το ταμείο αυτό ε, δεν παίρνουμε τα υπολείμματα των άλλων ταμείων, το παίρνουμε από τη μία κοινωνική τσέπη και τα πάμε στην άλλη. Ε, πρέπει να το ξέρουμε αυτό στο μέλλον. Τώρα οι εγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις μέχρι στιγμής σας το είπα ήταν πολύ γενναιόδορες ε, και λόγω της ε, αυστηρής στάσης του Προέδρου μας που ζήτησε δεν επέτρεψε, μου συγχωρείτε, κάποιε βελτιώσει. Δεν ήταν καλά δομημένε και δεν ήταν και καλά αποτελεσματικέ, κατά την άποψή μου. Οπότε, εγώ θα ήθελα οπωσδήποτε κάνουμε το καλό, αλλά πρέπει να βοηθάμε και σε βάθος χρόνου. Οι πολίτες, κύριε Πρόεδρε, από εμά δεν αναμένουν μόνο να ανοίγουμε την κάνουλα και να μοιράζουμε λεφτά, αλλά αναμένουν να το κάνουμε και κάπως λογικά. Είναι τα δικά τους λεφτά που μοιράζουμε. Και πρόθεσή μου είναι πραγματικά να τα χρησιμοποιούμε αυτά λογικά. Και υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα προς αυτή την κατεύθυνση με το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Στάουνερ και τώρα για την ε, προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών ε, για αυτόν τον κανονισμό την έχουμε ορίσει στις 13 Φεβρουαρίου έως τις 12 το μεσημέρι λίγη το θέμα. Πάμε στο επόμενο σημείο της κυρίας Μαντέιρα. για την υγεία και την ασφάλεια, για τις ε, εγγύους, για τις λεχόνες. Κυρία Μαντέιρα, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Ευχαριστώ όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου για την ε, συζήτηση πριν από την πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή. Ε, πολύ χρήσιμη η συνεισφορά τους. Ε, πρόκειται για μια τροποποίηση του κανονισμού ε, ε, που έχει ένα καινοτόμο στοιχείο, δηλαδή επιτρέπει με κάποια μορφή την την εφαρμογή της αρχής ε, ε της ε, ίσης μεταχείρισης ανάμεσα άντρες και γυναίκες βάσει το 170, άρθρο 171 της ε, συνθήκης και πραγματευόμαστε την ισότητα στην αγορά εργασίας και η πρότασή μας που αναπτύσσουμε μέσα σε αυτή την γνωμοδότηση Κυρία Στάουνερ και ο βοηθός σας, σας παρακαλούμε πάρα πολύ λίγη ησυχία. Ε, έλεγε λοιπόν η κυρία Μαντέιρα ότι πραγματευόμαστε αυτή την ε, πρόταση μέσα στο σχέδιο χνομοδότηση, ώστε η γυναίκα να έχει την ε, δυνατότητα να κάνει τις επιλογές για τη ζωή της. Τι εννοώ η μητρότητα είναι χαρακτηριστικό των γυναικών. Εντάξει, αυτό είναι στοιχείο κλειδί, τι να πούμε. και μιλάμε για την ε, προσωπική ανάπτυξη, για την ε, συμφιλίωση της ε, ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Είναι οι τρεις πυλώνες και που δεν συνδυάζονται ορισμένε φορέ. Ορισμένοι παρετούνται από την επαγγελματική του ζωή, από την οικογενειακή ζωή, από την ιδιωτική και από τα δύο. Τέλο πάντων, υπάρχει ένα ανταγωνισμό ανάμεσα σε αυτέ τι τρει συνιστώσει. Μα αυτό δεν είναι ο στόχο μα, ούτε και είναι ο στόχο μα. Όταν μιλάμε ειδικά για τις γυναίκες και για το δικαίωμά τους να γίνουν μητέρες. Γιατί για την πρόσβαση στην αγορά εργασία ε, με την τωρινή κατάσταση πλήγονται περισσότερο οι γυναίκες. Και δεν μιλάμε μόνο για την πρόσβαση, μιλάμε και για την παραμονή τους ε, στην αγορά εργασία. Οπότε ε, θέλουμε να κατοχυρώσουμε θα κάνει επιλογές η γυναίκα σε ασφαλείς, υπό ασφαλείς συνθήκες και εγγυόμενη και την ασφάλεια αλλά και την υγεία των εργαζομένων θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό γιατί δεν έχουμε μόνο τη σωματική, έχουμε και την ε, ψυχική υγεία. Ε, και σε κάθε προσωπική επιλογή ε, αν υπάρχει οποιαδήποτε αντικσότητα πλήττεται και η σωματική και η ψυχική υγεία. Τώρα μιλάμε για την άδεια της μητρότητας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα συμφιλίωσης των απόψεων. Υπάρχει το θέμα της οδηγίας της γονικής άδειας, που είναι άλλο ξεχωριστό θέμα, και η οδηγία για τους αυτοαπασχολούμενους. Και δεν αγγίζουν μόνο αυτά τα ζητήματα, αλλά αγγίζουν και αυτό το θέμα της ε, άδειας της ε, μητρότητας, αλλά και της πατρότητας. Ε, θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία στην κατανομή των ευθυνών. Αυτό είναι το βασικό κόλλημα για να υπάρξει αυτή η ισορροπία ανάμεσα στους τρεις πυλώνες ε, ε, και να κατοχυρώνεται η ελευθερία της επιλογής. Γι' αυτό δεν εκπληρώνει το στόχος, γι' αυτό δεν επιτυχάνεται η ισορροπία ανάμεσα στις τρεις αυτές συνιστώσεις. Θέλουμε να περάσουμε από τους 14 28 εβδομάδες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι 6 υποχρεωτικές εβδομάδες. Πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία της πρότασης Επιτροπής ε, και συγκεκριμένα θέλω να τονίσω το θέμα της ευθύνης. Ε, στην ευρωπαϊκή ευθύνη. Μιλάμε για την γύρανση του πληθυσμού και για τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η μητρότητα, ο κοινωνικός ρόλος των γυναικών, η άσκηση του δικαιώματα στους να γίνουν μητέρες. Σας μίλησα για αυτές τις τρεις συνιστώσεις, ε, αλλά δεν πρέπει αυτό να επηρεάζει την επιλογή της γυναίκας να χρειάζεται να παρετείται από αυτό το δικαίωμά της. Χρειάζεται να, ε, να θεσμοθετήσουμε εργαλεία που θα ε, διαφυλάξουν τα ε, δικαιώματά της. Είπαμε ότι περνάμε τους 6 12 μήνες για την απαγόρευση απόλυσης. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Γιατί Ακόμη και όταν μιλάμε για τον άλλο γονιό, για τον πατέρα δηλαδή, ε, όταν ε, έρχεται ένα παιδί στο σπίτι, ανα, αναταράσσεται η ισορροπία στο σπίτι, αναδιοργανώνεται το σπίτι και η οικογενειακή ζωή. οι 18 εβδομάδες για την επιστροφή της γυναίκας στην αγορά εργασία. τι σημαίνει αυτό. Όχι μόνο πρέπει να αναδιοργανωθεί στην προσωπική ζωή, αλλά και στην επαγγελματική. Χρειάζεται να διοργάνωση λοιπόν τη επαγγελματική ζωή και στα, στις διάφορες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θυλασμό αυτή είναι η περίοδος αναφοράς, αν θέλετε, που συστήνουν οι γιατροί, έξι μήνες για το θυλασμό. Και ξέρετε ότι μπορεί αυτό να λειτουργήσει εις βάρος της γυναίκας. Ε, αυτοί οι έξι μήνες μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο απαιτούμενος χρόνος αλλά μπορεί να χρειαστεί και περισσότερος ε, χρόνος ε, για την αποκατάσταση της ε, κανονικής ζωής, για να καταφέρει δηλαδή οι εργαζόμενοι προκειμένου να ανταπεξέλθει. Όταν τώρα για μία έγκυο υπάρχει αυτή η ανάγκη τη ε, της ε, κοινωνική ασφάλισης, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως ε, αλλαγή στη θέση εργασίας, νυχτερινή εργασία και οτιδήποτε άλλο. Άλλε ειδικέ ανάγκες θα πρέπει να καλύψουμε και αυτή την περίπτωση. Βέβαια υπάρχουν ρυθμίσεις σε άλλα νομοθετήματα, αλλά ξέρουμε πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας και έχει ιδιαίτερη σημασία να το ρυθμίσουμε και αυτό, ούτως ώστε να μην υφίστανται διακριτική μεταχείριση ή οσδήποτε μορφή οι γυναίκες ε, στην αγορά εργασίας. Μετά τις 18 εβδομάδες ε, που λείπουν από την αγορά εργασίας, οι εργαζόμενες ε, και ξέρετε πόσο ευμετάβλητο είναι το κλίμα στην αγορά εργασίας. Η παραγωγική διαδικασία, τώρα ειδικά με την ε, οικονομική κρίση, και πολύ καλό που την κάνουμε τώρα τη συζήτηση και όχι νωρίτερα, οι 18 εβδομάδες σημαίνουν μπορεί να είναι επίκαιρες πλέον οι δεξιότητες της εργαζόμενης σε σχέση με τις προοπτικές της, τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές ε, μετά τον τοκετό. Άρα, χρειάζεται να προβλέψουμε κατάρτιση, επιπλέον κατάρτιση, ούτω ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει η εργαζόμενη όταν θα επιστρέψει μετά τον τοκετό. Αν τυχόν και αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ε, ο μισθός κατά την ε, άδεια της μητρότητας, να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνούμε απολύτως με τις προτάσεις Επιτροπής. Και πέρα από τη διατήρηση του εισοδήματος του μισθού, πρέπει να υπάρχει και άλλο ηχέγγυο ότι δεν θα πληγούν τα συνταξιδοτικά συστήματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συντάξεις και διαφορετικές ερμηνείες, αλλά Επίσης, ε, ε, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου της άδειας ε, πρέπει να κατοχυρωθούν και τα συνταξιδιωτικά δικαιώματα για να αντιμετωπιστεί το θέμα, το πρόβλημα της ευτόχειας μετά το τεπέρας της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πρέπει να θωρακιστούν και αυτά τα δικαιώματα. Το θέμα της κατανομής των ευθυνών είναι δύσκολο πέρα από το θέμα της νομικής βάσης που συνεχίζει να τίθεται. Ε, η Επιτροπή τι μας λέει. Ε, ο εργοδότης ε, να είναι υποχρεωμένος να εξετάζει το αίτημα για την αλλαγή των ωραρίων χωρίς αυτό να είναι έκτακτο μέτρο, να είναι ε, τακτικό μέτρο. Ε, είτε υποβάλλει το αίτημα ε, η μητέρα, ο πατέρας, ο σύντροφος, όλα εν πάση περιπτώσει τα τεινά που συμβαίνουν ω προ τη συμβίωση, όποιο και να είναι που εντάσσεται στα, στα, πλαίσια, δηλαδή οποιοδήποτε από το ζευγάρι υποβάλλει την ε, αίτηση, θα πρέπει να υποχρεώται ο εργαδό να την εξετάσει. Αυτό για να συμφιλειωθεί η οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Τώρα για του αυτοαπασχολούμενου. Όπω έλεγα στην αρχή, ε, ε, δεν είναι ο στόχος ο βασικός της οδηγίας, αλλά είναι δίκαιο να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της Επιτροπής μας. Γι' αυτό προτείνω νέο άρθρο 9, ούτως ώστε ανεξάρτητα από τις τροποποιήσεις ε, της οικίας εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να μεριμνήσουν όλα τα κράτη-μέλη να ε, μεριμνήσουν και για τους αυτοαπασχολούμενους είναι ένα πολιτικό μήνυμα ε, και μόνο, αλλά τέλος πάντων έχει αυτή την αξία του. Και κάθε κράτος μέλος θα το ερμηνεύσει ε, όπως καταλαβαίνει αυτό το πολιτικό μήνυμα. Θα κλείσω σε λίγο. Απλά ήθελα να τονίσω ότι για την υγεία, θέμα της υγείας, υπάρχει μία σύσταση από το 2002 που αναφέρεται στην διατροφή του νηπίου, του βρέφους. Κατά τη διάρκεια των, του θυλασμού, τους πρώτους έξι μήνες. Για μας είναι πολύ σημαντικό το θέμα του θυλασμού αυτούς τους πρώτους έξι μήνες. Προτείνεται εδώ αν η μητέρα επιλέξει το θυλασμό, να προσθεθούν άλλες έξι εβδομάδες. Από 20... Να γίνουν 24 εβδομάδες της άδεια μητρότητας, δηλαδή αν ε, θυλάσει η μητέρα. Είναι σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι άλλο ξέχασα να σου πω κάτι στην αρχή, αλλά τέλος πάντων είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό το πω τώρα. Μιλήσαμε για την άδεια μητρότητας και εμπλέκονται διάφορες οδηγίες, αλλά ε, μην ξεχνάμε τα μήνυμα, τα μήνυμα των στόχων της τις ε, της διαδικασίας της Βαρκελόνης για την υποστήριξη της οικογένειας ε, και των παιδιών. Συμβαστικές λύσεις, οι οποίες έχουν καταλήξει τα κράτη-μέλη, πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους σε σχέση με αυτές τις δεσμεύσεις και για να εκπληρώσει το στόχο της ε, η οδηγία θα πρέπει να ξαναφέρουμε στο φως της ημέρας αυτές τις δεσμεύσεις που ήδη έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη. Πολύ σας ευχαριστούμε. Τρεις έχουν, ε, θέλουν να μιλήσουν, η κυρία Στάνερ και η κυρία Λίν αρχικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεγέτρια, είπατε ότι η μητρότητα ε, συνδέεται άρρηκτα με την ύπαρξη της γυναίκας. Είναι σωστό. Αλλά δυστυχώς ε, γνωρίζουμε ότι ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σύνηθες πλέον εν γέννη κάθε γυναίκα να αποκτάει παιδιά. Και νομίζω ότι θα έπρεπε πραγματικά να φροντίσουμε ούτως ώστε η περίοδος που οι γυναίκες απομακρύνουν από την εργασία τους επειδή έχουν αποκτήσει ένα παιδί κατά κανένα τρόπο να μην προσλαμβάνεται σαν ένα μειονέκτημα. Είμαι απόλυτα σύμφωνη με την ε, αύξηση από 14 σε 18 εβδομάδες της προθεσμίας. Αλλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες που ούτως ή άλλως υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το όριο μέχρι τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια την άδεια δηλαδή όχι μόνο υπό την έννοια της μεταχείρισης Δηλαδή όχι μόνο υπάρχουν ε, αυτά τα διαστήματα, δεν προβλέπονται μόνο για τις μητέρες αλλά και για τους πατεράδες. Είναι και στην Κομισιόν υπάρχει προβληματική ότι δεν είναι μόνο οι εργαζόμενες γυναίκες ή οι εργαζόμενοι γονείς που επιθυμούν να επιστρέψουν στην εργασία τους το δυνατό μετά την γέννηση του παιδιού, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι γονείς που θέλουν να αναθρέψουν μόνοι τους τα παιδιά. Ε, δηλαδή ένας πατέρας ή μία μητέρα και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η Κομισιόν προτείνει ένα υποχρεωτικό διάστημα έξι εβδομάδων μετά τον τοκετό και διαρωτώμε κατά πόσο δεν θα είχε νόημα πριν από τον τοκετό να θεωρηθεί υποχρεωτικό ένα χρονικό διάστημα άδειας της μητέρας γιατί αν το ότι γίνεται στις πιο επισφαλείς συνθήκες εργασίας ε, μπορώ να φανταστώ ότι αν δοθεί άδεια στο χρονικό διάστημα πριν από το κετό τότε οι εργοδότες ε, θα ασκήσουν ε, πίεση στις μητέρες να εργάζονται μέχρι τη στιγμή του τοκετού. Όσον αφορά την προθεσμία ε, βλέπω τον κίνδυνο. Εάν περάσει αυτή η προθεσμία με την τελευταία ημέρα της ε, προθεσμίας που προβλέπεται για την άδεια μητρότητας, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα για τη γυναίκα. Διότι όταν επιστρέψει η γυναίκα στην εργασία της θα ανακύψουν ενδεχομένω κάποια προβλήματα, δηλαδή θα μπορεί να είναι έγκαιρα στην, στο χώρο εργασία κλπ. Θα πρέπει λοιπόν η προστασία αυτή έναντι των επολύσεων θα πρέπει να ξεπερνάει το διάστημα της άδεια μητρότητας, η προστασία έναντι των απολύσεων. Γιατί και εκεί μπορεί η γυναίκα να μην είναι απολύτω συνεπή προ τη δουλειά τη. Τώρα, η συγγήτρια κατέθεσε μια ε, τροπολογία ε, όπου λέει ότι το να μην ε, εξαλείψει κανείς την άδεια μητρότητας δεν θα πρέπει ε, το να, συγγνώμη, να έχει ε, μια γυναίκα την άδεια μητρότητας αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρνητική επίπτωση στη σταδιοδρομία της γυναίκας. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το εκφράσουμε αρνητικά, αλλά με θετικούς όρους. Θα πρέπει να πούμε ότι η άδεια μητρότητας επηρεάζει θετικά την ε, σταδιοδρομία της γυναίκας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να, κάνουμε, να προσπαθούμε να προστατεύσουμε γυναίκες απλώς και μόνο επειδή θέλουν να εργάζονται και να είναι ταυτόχρονα και μητέρες. Δεν χρειάζεται μια επιπλέον προστασία δηλαδή. Κυρία Λίν. Ευχαριστώ. Θα Ε, δεν πρέπει εδώ να δίνουμε την εντύπωση ότι λέμε στις γυναίκες ότι οπωσδήποτε πρέπει να λείψετε έξι εβδομάδες. Εκείνες θα τα αποφασίσουν. Οι ενδιαφερόμενες εμείς η Ένωση ή οποιοδήποτε άλλος θα τους επιβάλλει ότι ντε και καλά ε, υποχρεωτικά πρέπει να ε, μείνει στο σπίτι ε, έξι έξι μήνε ή, εν πάση περιπτώσει, άμα θέλει να γυρίσει νωρίτερα ή άμα θέλει να δουλεύει μέχρι τελευταία στιγμή, δικαίωμά τη είναι. Δεν μπορούμε να το, τους το επιβάλλουμε. Δηλαδή, αυτή η υποχρεωτικότητα της άδεια με αφήνει αναβδί. Και αυτά που είπατε στην αρχή της παρέμβασής σας ε, για την, ε, ε, τον επιμερισμό της άδειας, άδεια μητρότητας και πατρότητας, Καλά λέτε ότι πρέπει να εξετάσουμε από κοινού όλες εμπλεκόμενες οδηγίες. Οι γονεί ε, συνήθως αποφασίζουν μεταξύ τους ε, ποιος θα φροντίσει το παιδί, ποιος θα μείνει με το παιδί. Αν θέλει ο πατέρας, ε, πολλέ φορέ θα αποφασίζει να παραμείνει αμέσως μετά το τοκετό με το παιδί. Σε άλλες περιπτώσεις η μητέρα αποφασίζει να παραμείνει με το παιδί. Τέλος πάντων, για τον επιμερισμό των ευθυνών, εγώ πιστεύω ε, θέρμος ότι τα ίδια δικαιώματα έχουν και οι πατέρες μπορεί για να αποκτήσουν στενή σχέση με τη μητέρα. Για την ε, προστασία από τις απολύσεις. Αν ε, το τραβήξουμε ακόμη περισσότερο θα έχουμε πολύ περισσότερες προσφυγές στο δικαστήριο. Δηλαδή θα πούνε κάποια, δεν μπορώ να επανέλθω στην αγορά εργασία γιατί δεν έχω πλέον τι απαιτούμενε δεξιότητε. Καμία σχέση με την εγκυμοσύνη αυτό. Για τους αυτοαπασχολούμενους τώρα. Καλή ιδέα να τους ε, καλύψουμε, αλλά πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Ε, θα ήθελα να το εξετάσουμε με περαιτέρω. Εμείς έχουμε και μισθό κατά την άδεια της μητρότητας και επίδομα την, ε, για τη μητρότητα. Ε, το επίδομα είναι άμα δεν ε, δουλεύατε όταν μείνατε έγκυος παραδείγματος χάρη και αυτό γίνεται με τις κοινωνικές εισφορές, έτσι χρηματοδοτείται. Τώρα, εάν είστε αυτοπασχολούμενοι και γεννήσετε πρέπει να πληρώσει οι αυτοπασχολούμενοι υψηλότερες κοινωνικές ε, εισφορές ε, ενώ στην αντίθετη περίπτωση μια μισθωτή όχι για να καλυφθεί το επίδομα μητρότητας. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Πώς, τι θα γίνει με το επίδομα μητρότητας και το μισθό κατά τη διάρκεια ε, της ε, ε, άδειας μητρότητας. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό για τους αυτοαπασχολούμενους. εφόσον ε, οι αυτοαπασχολούμενοι επιλέγουν πότε θα δουλέψουν και πότε θα δουλέψουν, θα πούνε οι άλλοι γιατί να πληρώνουμε εμεί τα σπασμένα για αυτού. Ε, μπορούν οι ίδιοι να πάρουν την άδεια τη ε, μητρότητα και να την πληρώσουν μόνοι του. Εγώ δεν είμαι κατά του να συμπεριλάβουμε τους αυτοπασχολούμενους, αλλά δεν καταλαβαίνω στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Νομικός πώς το, τα κράτη-μέλη μπορούν να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους για να ευθυγραμμιστούν με τις νέες διατάξεις. Νομίζω θα δημιουργηθούν πολλά πρακτικά προβλήματα. Τα είπα για τις υποχρεωτικές έξι εβδομάδες, τώρα θα σας πω για τη μη υποχρεωτική περίοδος, οποιαδήποτε στιγμή μείνει έγκυος μία γυναίκα. Άλλο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, γιατί πώς θα ελέγξουν το εργατικό τους δυναμικό Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να την πάρει την άδεια η γυναίκα, ε, θα είναι πρόβλημα αυτό για τις επιχειρήσεις, για κάποιες από τις επιχειρήσεις. Ε, πρέπει να βρούμε έναν ε, μηχανισμό για να δούμε πώς θα είναι εφικτό, πώς δεν θα πούνε οι επιχειρήσεις όπως και στο παρελθόν ότι ε, λοιπόν εμείς δεν θα απασχολούμε κάποιες γυναίκες ε, και μιλάμε για νομοθεσία με στόχο την κατάρριξη της διακριτικής νομοθεσίας και αν δεν εμείς ε, δεν ε, ξασφαλίσουμε ισοτιμία ανάμεσα στα δικαιώματα του πατέρα και της μητέρας, ε, θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Κάποιες γυναίκες κάποιας ηλικία δεν θα βρίσκουν δουλειά. Γιατί ακριβώς είναι αυτή τη ηλικία. Κατοχυρώσουμε λοιπόν ταυτόχρονα με τα δικαιώματα της μητέρας και τα δικαιώματα του πατέρα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σρέτερ και η κυρία Πλάν. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά η προσέγγιση και η τροπολογία της κυρίας Μαντέρα είναι σωστές και τα υποστηρίζουμε. Αυτό το οποίο είναι προβληματικό για εμένα είναι το ζήτημα το να μπερδεύουμε την άδεια την ε, γονεϊκή με την μητρότητα γιατί η μητρότητα είναι ζήτημα και προστασία στην ε, εργασία και αφορά και τις γυναίκες που είναι μόνες τους και εδώ πέρα μιλάμε προστασία ε, της υγείας των γυναικών που είναι μόνες τους και πρέπει να δουλέψουν για να αναθρέψουν το παιδί τους και αυτό σημαίνει ναι, έχουμε γονείς, έχουμε μάλλον ε, την ε, γονική άδεια που αναφέρεται σε άλλη οδηγία, ίσως και καλύτερα, σε αυτό είμαι ανοιχτή, αλλά ποια είναι η δυσκολία. Είναι αν ρυθμίζεται καλά στα κράτη-μέλη, μήπως είναι σε χειρότερη θέση μάλλον οι γυναίκες οι οποίες αναθρέφουν μόνες τους το παιδί τους. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Κομισιόν να μας πει έφερε αυτή την, ε, την τροπολογία γιατί θέλει να προστατεύσει καλύτερα τις γυναίκες ακριβώς εκείνες οι οποίες πρέπει να επανέλθουν στη, στην εργασία τους για να δούμε και αυτούς τους 6 με, με 12 μήνες για να διορθωθεί αυτή η ανισότητα. Την υποστηρίζουμε αυτή την τροπολογία αλλά δεν ξέρω εάν είναι σωστή αυτή η σύγχυση που, που γίνεται και αν ισχύει αυτό για τις ε, γυναίκες εάν είναι μόνες τους ή όχι και αν ισχύει για όλες τις ε, γυναίκες που πρέπει να, να προστατευτούν. Και το ερώτημα βεβαίω πότε θα λάβουν αυτή την, την άδεια ή τις μέρες αυτές και πώς και τα λοιπά γιατί υπάρχουν ε, και διαφορετικές ε, καταστάσεις ε, και το πώς αισθάνεται η γυναίκα στη μία στην άλλη φάση. Γι' αυτό θεωρώ σωστή εδώ πέρα την πρόταση της ε, Κομισιόν που είναι ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Επίσης το θέμα της περαιτέρω κατάρτισης γιατί πράγματι υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει μετά να επανέλθει στην ίδια εργασία. Τώρα, όμως η προσθήκη εδώ στην τροπολογία 10 καθιστά πιο ανίσχυρο το... τη διατύπωση αυτή. Καλύτερα να τα αφήσουμε όπως το έχει η Κομισιόν, να μην τον ερώσουμε. Θα ήμουν πιο προσεκτική Πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι και να μην το νερώσουμε, να μην το αποδυναμώσουμε. Πέρα αυτά από μένα. Η κυρία Πλούμ και η κυρία Τόμασεύσκα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Μαδέρα για την έκθεσή της. Είμαι απολύτως σύμφωνη με την έκθεσή της και θα ήθελα να πω ότι στηρίζω όλες τις ε, βελτιώσεις που επιφέρει στην οδηγία μέσω της έκθεσής της. Θα ήθελα να σας πω ότι υποστηρίζω την ιδέα να αυξηθεί η άδεια μητρότητας μέχρι τις 24 εβδομάδες και αυτό για δύο λόγους. Καταρχήν, πρόκειται εδώ για την φυσική εκπαίδευση, τη συλλογική εξέλιξη του παιδιού. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν αυξήσουμε μόνο κατά τέσσερις εβδομάδες αυτή την περίοδο σε σχέση με τη μητρική άδεια, κάτι που ε, ήδη εφαρμόζουν στην πράξη αρκετές χώρες μέλη, τελικά δεν θα σημειώσουμε ιδιαίτερα μεγάλη πρόοδο. Η εφαρμογή της οδηγίας θα γίνει μέσα σε δύο χρόνια από την έγκρισή της. Το δεύτερο πρόβλημα ε, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εξή. Πρόκειται για τις απολύσεις. Στο πρωταθέν από την Επιτροπή κείμενο αναφέρεται το ότι ο εργοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει γραπτά εύλογα επιχειρήματα για την απόλυση μιας γυναίκας εργαζόμενης. Πιστεύω ότι αυτοί οι τεκμηριωμένοι λόγοι θα πρέπει να διευκρινίζονται. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί προέρχομαι από τη Ρουμανία. Η επιθεώρηση εργασίας στο Εθνικό Συμβούλιο κατά των διακρίσεων και εδώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι ο εργοδότης για λόγους απολύτως, απολύτως δικαιολογημένος κατά την άποψή του διέκοψε το σύμβαση εργασίας της γυναίκας κατά τη διάρκεια της κοίησης ή το και του. Γι' αυτό εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση αυτής της έννοιας του καλώς τεκμηριωμένη λογη Κατά τα άλλα είμαι σύμφωνη για τις τροπολογίες που κατατέθησαν από την κυρία Μαϊδέρα και θα ήθελα να επαναλάβω ότι την υποστηρίζω πλήρως. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Τόμασεύσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ζητήματα θα ήθελα να θίξω. Το πρώτο αφορά αυτό το οποίο η κυρία Λίν για τους μηχανισμούς, για το πώς θα πληρώσουμε τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά ταμεία που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως του, της εργασιακής του σχέσης. Φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και το πώς θα οργανωθεί. Υπάρχει εδώ πέρα μια κοινωνική αδικία γιατί οι γυναίκες που έχουν παιδιά γιατί οι γυναίκες δεν, αυτές δεν μπορούν να εργαστούν για αρκετά μεγάλο διάστημα, δεν έχουν χρήματα ή έχουν τόσο κάποια χρήματα αναλόγως με το που ζουν και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα τους και στο μέλλον έχουν μικρότερη σύνταξη. Αλλά τα παιδιά τους, λόγω της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, ε, που θα πληρώσουν ε, ούτως ή άλλως αυτές τις εισφορές τις παραπάνω για τις γυναίκες που δεν έχουν κάνει παιδιά. Και για αυτές μάλλον. Οπότε είναι κάτι το οποίο απαιτεί ειδικού μηχανισμούς. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο ζήτημα Γιατί είναι γυναίκες που γεννάνε νωρίτερα και είναι υγιέστερα τα παιδιά και είναι... Τα παιδιά που θυλάζουν είναι πολύ πιο ανθεκτικά στις ε, ασθένειες, έχουν καλύτερο ανασωπητικό κλπ. Γι' αυτό θέλω να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Έχει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση που περιέχει πολύ σημαντικά ερευθίσματα και αναφέρεται πολύ λεπτόμερο στην πρόταση. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε όλες τις τροπολογίες, κάποια πραγματάκια μόνο να υπενθυμίσω που μου φαίνονται κάπως σημαντικά. Στην πρόταση ε, έχουμε δύο νομικές βάσεις το 137 και το 141 έχουμε αυτά τα δύο άρθρα γιατί αφενός έχουμε κατά νου την υγεία της μητέρας δηλαδή την πτυχή υγείας και ασφάλειας και αφετέρου την πτυχή του να συμφιλιώσουμε την εργασία και την οικογένεια και θέλουμε να το ενισχύσουμε αυτό. Δηλαδή να λέμε ότι δεν πρόκειται μόνο για την υγεία και την ασφάλεια, εντάξει σε μεγάλο βαθμό οπωσδήποτε, αλλά έχουμε και την πτυχή συμφιλίωσης αυτής υγείας και οικογένειας. Γι' αυτό ε, ενισχύσαμε τον ρόλο των γυναικών με πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας και κάπως περισσότερο. Και κάποια άλλα πράγματα. Επίσης ε, συζητήθηκε στην Επιτροπή Γυναικών το να μην αναφερθούν ρητά οι πατεράδες. Θέλω να το αναφέρω. Δεν συμπεριλάβαμε τους πατεράδες γιατί θεωρούμε πως η νομική βάση εδώ πέρα δεν μας καλύπτει για κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα μιλάμε για τροποποίηση μιας οδηγίας 1997 και θεωρούμε πως ε, δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα ξαφνικά τους πατεράδες αν και βεβαίως υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα και ελπίζουμε πως οι κοινωνικοί εταίροι στους διαπραγματεύσεις θα μιλάνε για γονείς και για τους δύο γονείς άρα θα συμπεριλάβουν ένα τέτοιο δικαίωμα. Εάν δεν γίνει αυτό, οπωσδήποτε θα πρέπει να τοποθετηθεί η Κομισιόν, αλλά είναι σαφές πως η Κομισιόν συνολικά είναι πολύ θετική να επεκταθεί αυτό το, το δικαίωμα. Ούτως ή άλλως το δικαίωμα της ε, άδειας πατρότητας αναφέρεται σε πολλές οδηγίες και γνωρίζει γενικότερα τι στάση μας, αλλά όπως σας είπα η αιτία είναι ε, η νομική βάση που θεωρούμε ότι δεν, δεν μας στηρίζει. Το ίδιο ισχύει και για αναφορές που γίνονται για τους γονείς διαχωρίσαμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε το δικαίωμα και τον αυτοαπασχολούμενο το οποίο δεν συμπεριελήφθη γιατί αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε μια αλλαγή σε μια οδηγία που θα δημοσιευτεί ταυτόχρονα με αυτήν εδώ την πρόταση. Η 82378 η οδηγία που θα ξεκαθαρίσει αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό δεν το συμπεριλάβαμε σε αυτή την οδηγία, αλλά σε μια άλλη, γιατί είναι ελαφρώς διαφορετικό το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό απασχολούμενοι οπωσδήποτε δεν ε, μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να πάρουν ε, άδεια μετρώτα... Το ξέρουν οι ίδιοι και το κανονίζουν. Εάν και αν θέλουν βεβαίως να σκίσουν αυτό το δικαίωμα δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό. Οπότε το αφήνουμε κατά μέρος αυτό το, το πρόβλημα και θα α, μας απασχολήσει σε άλλη οδηγία. Κατά τα άλλα, να υποστηρίξω αυτό το οποίο ήδη ακούστηκε στην Επιτροπή. Πράγματι, το θέμα εδώ πέρα αφορά και τις μόνες μητέρες που δεν μπορούν οπωσδήποτε να εκμεταλλευτούν αυτή την άδεια γιατί δεν μπορούν να ζητήσουν να πληρωθούν ε, αυτή τη γονική άδεια. Και σε πάρα πολλά κράτη-μέλη η γονική άδεια είτε δεν πληρώνεται είτε πληρώνεται ελάχιστα. Γι' αυτό οι γυναίκες οι οποίες είναι μόνες τους πρέπει πράγματι να έχουν δικαίωμα σε γονική άδεια που θα πληρώνεται για να έχουν καλές συνθήκες και αυτές για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους όταν μεγαλώσει κάπως το, το παιδί τους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας μήνας, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και βεβαίως με τις οδηγίες ε, ως γνωστόν ορίζουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις και όχι τις μέγιστες απαιτήσεις και θεωρούν πως με αυτές τις 18 εβδομάδες ε, επιτύχαμε κάτι το οποίο είναι επιτεύξιμο και ανταποκρίνεται σε αυτό το χαρακτήρα των ελαχίστων όπως ε, σα είπα και τηρήσαμε αυτό το οποίο είναι ο κανόνα σε πολλά κρατημέλη πολλά κρατημέλη έχουν αυτούς 18, 18 εβδομάδες αναφέρεται σε μια σύσταση του διεθνού Οργανισμού εργασία, Διεθνού Γραφείου εργασία. Προσπαθήσαμε δηλαδή να βρούμε μια βάση το δυνατόν πιο γενικά αποδεκτή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 που μίλησαν για την έκθεση και για την πρόταση της Επιτροπής. Πριν κάνω κάποια σχόλια, θα ήθελα να ρωτήσω αν δεν, έχει, δεν θέλει να τοποθετεί το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Δεν είναι εδώ. Ωραία λοιπόν, δεν παρευρίσκεται το Συμβούλιο. Ωραία λοιπόν, Τώρα θα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σχόλια και σε ορισμένες ε, ε, από ορισμένες παρεμβάσεις μπορώ να κρίνω ότι προχωρούμε όλοι στην ίδια γραμμή. Ε, το ζήτημα των εβδομάδων να δίδεται άδεια πριν από την ημερομηνία του τοκετού. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στην πρόταση τη οδηγία. Να δίδεται άδεια δηλαδή πριν από τον τοκετό και όχι μόνο μετά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντοτε εξετάζουμε από δύο οπτικές γωνίες, γιατί μπορεί ενδεχομένως να ζημιώσει την ε, δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης της γυναίκας μετά το τοκετό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την άλλη ε, σε περίπτωση που υπάρχουν κίνδυνοι στην εγκυμοσύνη. Και ίσως στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης θα μπορούσε να φροντίσει να πάρει κανείς την άδεια μικρότητας νωρίτερα. Να πάρει μια γυναίκα την άδεια μικρότητας νωρίτερα. Υπάρχουν πολλά υπέρ και κατά. Ε, δεν είναι εύκολο να τα ζυγίσει κανείς. Αλλά εμείς είμαστε υπέρ η γυναίκα να έχει η ίδια την εκλογή, εφόσον το επιθυμεί, να πάρει την άδεια αυτή μία εβδομάδα νωρίτερα, ούτω ώστε να προστατευτεί από τους τυχόν κινδύνους που επιφέρει ένας τοκετός. Εγώ μίλησα με νοσοκόμες, με ορισμένες ΜΕΣ και όλοι μου είπαν ότι ενδεχομένω μία ή δύο εβδομάδες πριν από το κοιτό ενδείκνυται, αλλά ενδεχομένω και ένας μήνας σύμφωνα με ορισμένους. Όλα αυτά, ε, όλες τις προτάσεις στηρίζουν σε κάποια επιχειρήματα. Θα πρέπει η δυο εβδομαδε πριν απο το κοιτο ενδεικνυται αλλα ενδεχομενω και ενα μηνα συμφωνα με ορισμενου ολα αυτα ολες τι προτασεις στηριζουν σε καποια επιχειρηματα θα πρεπει η γυναίκα να μπορεί να το κρίνει και να το αξιολογήσει. Ε, υπάρχει το επιχείρημα ότι η γυναίκα παίρνει αναρωτική άδεια στην περίπτωση αυτή πριν από τον τοκετό και αυτό δεν είναι επιθυμητό. Όσον αφορά τις αυτοπασχολούμενες, βεβαίως αυτό είναι ένα εντελώς ξεχωριστό σύστημα. εάν πραγματικά και 27 χώρες μέλη έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κατοχυρώσουν τις γυναίκες, ε, τα πράγματα θα είχαν καλώς. Αλλά όπως βλέπουμε υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας κλπ. κλπ. Και όπως σας είπα για τις αυτοπασχολούμενες ε, γυναίκες, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και πολύπλοκα. Ε, το άρθρο αυτό θα μπορούσε ενδεχομένω να εξελιχθεί περισσότερο δηλαδή να κάνει κανείς την προσπάθεια να εφαρμοστεί το πνεύμα της οδηγίας στις χώρες μέλη πριν υποβάλει τη δική της πρόταση η Επιτροπή και να εφαρμοστεί και για τις αυτοπασχολούμενες. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ίση μεταχείριση στην αργόρα εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν διακριτά, διαφορετικά μέτρα, διαφορετικά συστήματα από χώρα σε χώρα και υπάρχουν και διαφορετικές εισφορές από χώρα σε χώρα ή υπάρχουν ε, συστήματα τα οποία είναι φορείς που είναι ιδιωτικοί, υπάρχουν άλλοι που είναι φορείς του δημοσίου κλπ. Βλέπουμε λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις στις διάφορες χώρες μέλη, αλλά το δικαίωμα επιλογής εκ μέρους της γυναίκες αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Όπως σας είπα, η γυναίκα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παίρνει την άδεια μητρότητας και αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να έχουν και οι αυτοπασχολούμενες γυναίκες. Και ε, αυτό είναι επιθυμητό και θα πρέπει να καθίσταται και εφικτό για όλες τις γυναίκες. Τώρα, εσείς με το όσα είπε η κυρία Σρότερ για αυτή την έκτακτη κατάσταση. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα της μετάφρασης. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Στην ε, πορτογαλική εκδοχή νομίζω ότι αποδίδεται ορθά είναι σωστή η μετάφραση. Εν ώψη ε, ε, της οικονομικής κρίσης, βεβαίως αναμενόμενα να κλείσουν πολλές επιχειρήσεις, να απολύονται οι εργαζόμενοι ε, και θα πρέπει να προσανατολιστούν προς μια άλλη απασχόληση. Και στην περίπτωση αυτή πλήττονται περισσότερο οι εργαζόμενες μητέρες και θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση τους, θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω ε, πώς είναι η γερμανική διατύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το σκεπτικό. Ότι οι γυναίκες που απομακρύνονται από το χώρο εργασίας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλωθούν στο ίδιο, ε, με τους ίδιους όρους όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι άλλες γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε και με αυτό το θέμα. 31 Φεβρουαρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τροπολογίες. 13 Φεβρουαρίου, με συγχωρείτε, βεβαίως 31 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει. Κατόπιν έχουμε μία μελέτη για τις ε, νέες μορφές ε, κινδύνων σωματικής και της ψυχοκοινωνικής υγείας στην εργασία. Έχουμε λοιπόν δύο μιλητές, τους κυρίους Μέουσεν και Χάουτμαν που θα μας κάνουν αυτή την παρουσίαση. Έχετε και τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω πως όταν κατέβηκε η οθόνη σταμάτησε εγκαίρως, οπότε ε, διατρέχετε κι εσείς αυτό τον κίνδυνο στην εργασία το να σε ορθώνει στο κεφάλι. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω την μελέτη μας για τους νέες μορφές σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας στην εργασία. Είμαστε Ρωτήσαμε ερευνητέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανού, Ολλανδού, Πολωνού, συναδέλφου από την Ισπανία, από την Ισπανία και την Πορτογαλία, οπότε είχαμε αρκετά κρατημέλη και περιφερειέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι Μέουσεν και η κυρία Χάουτμαν εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση και θα σα ε, παρουσιάσω γρήγορα την έκθεση, να σα δώσω τα βασικά σημεία και να πω λίγα πραγματάκια για τον πίνακα που είναι και στην σύνοψη που έχετε στις έκθεση και αν έχετε βεβαίως ερωτήσεις ή παρατηρήσεις παρακαλώ να με ρωτήσετε για να απαντήσουμε. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε εδώ πέρα 12 κινδύνους που έχουμε βρει που αυξάνονται και έχουμε τους, τις αιτίες αυτών των κινδύνων. Και παρατήρησα και στη συζήτησή σας, η παγκοσμιοποίηση προφανώς είναι ένας κίνδυνος. Εννοούμε βεβαίω την γρήγορη μετακίνηση εργαζομένων που προφανώς αυξάνει αυτούς τους κινδύνους στον χώρο της εργασίας. Τα δημογραφικά στοιχεία, σκεφτείτε τη γύρανση του εργατικού δυναμικού που είναι ένα ζήτημα που επίσης συζητάτε εδώ πέρα σκεφτείτε τους μετανάστες που πηγαίνουν και έρχονται στα κράτη-μέλη για να γεμίσουν τα κενά στην αγορά εργασίας και αυτό είναι ένας παράγον που προκαλεί αυτούς τους κινδύνους. Προφανώς η τεχνολογική καινοτομία. Βλέπετε στην έκθεσή μας πως περιγράφουμε τον κίνδυνο της ε, κινητικότητας της εργασίας λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στους υπολογιστές. Σαφώς αυτό επηρεάζει τους ε, κοινωνικούς κινδύνους στην εργασία και το όριο πλέον του να δουλεύει κανείς σε εταιρεία ή στο σπίτι του ε, είναι όλο και πιο δυσδιάκριτο. Επίσης έχουμε την αντίληψη των νέων κινδύνων, το πώς αντιλαμβάνεται κανείς αυτούς τους κινδύνους μεταξύ των πολιτών. Οι πολίτες λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν και μαζεύουν πληροφορίες από το ίντερνετ και αυτό βεβαίως ε, ε, μπαίνει και στο κοινωνικό διάλογο οπότε αποτελεί εδώ πέρα παράγοντα και βεβαίως υπάρχει αύξηση στους φυσικούς κινδύνους σκεφτείτε το SARS άλλες ε, λοιμώδεις ε, ασθένειες των ε, εργαζομένων π.χ. στα νοσοκομεία και αυτών που παρέχουν πρώτες βοήθειες. Οι κατηγορίες του κινδύνου είναι τέσσερις συνολικά. Μία φορά τις μειοσκελετικές διαταραχές που συνδυάζονται με την φυσική ακινησία και τους κινδύνους πολλαπλών παραγόντων, μετά έχουμε τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα, μετά έχουμε τις επικίνδυνες ουσίες, πιο παραδοσιακό ζήτημα, τα πιο συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή επικίνδυνες ουσίες, νέες τεχνολογίες και σωματικά ε, ζητήματα και τέλος έχουμε συγκεκριμένες ομάδες ε, στόχων, συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου. Και αυτό βεβαίως συνδέεται και με τους νέους κινδύνους που έχουμε εμείς βρει. Πρώτη ομάδα λοιπόν έχουμε τους νέους αυτούς κινδύνους σχετίζονται κυρίως με μειοσκελετικές διαταραχές επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ο κλάδος των υπηρεσιών αυξάνεται όπως μάλλον ξέρετε βλέπουμε πως ε, μειώνεται η, η σωματική δραστηριότητα στη δουλειά, πιο καθιστική η δουλειά με υπολογιστές και αυτό σαφώς επηρεάζει την υγεία των εργαζομένων. Αυτό είναι και το θέμα μας ε, και το βλέπετε αυτό και σε έναν άλλο κείμενο που έχουμε πριν ότι αυξάνεται και αφορά και τη δημόσια υγεία. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αυστηρή διάκριση ανάμεσα στη δημόσια υγεία και στους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Επίσης, ο τρόπος εργασίας, ο τρόπος ζωής στη δουλειά, δηλαδή υπάρχει κίνητρο να κινηθούν σωματικά οι εργαζόμενοι ή έχουν καθιστική δουλειά όλη μέρα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό σε βάθος χρόνου, επηρεάζει βεβαίως την κατάσταση. Παχυσαρκία είναι σαφώς ο κίνδυνος εδώ πέρα που παρουσιάζεται. Τέλος, την ομάδα αυτή το έχουν βρει και άλλες μελέτες. Έχουμε τις πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Ψυχοκοινωνικό βάρος συνδυασμένο με καθιστική εργασία και τα μειοσκελετικά που αναφέραμε μας δίνει πλέον παράπονα των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυτές τις συνθήκες πολύ περίπλοκα. Και αν βάλουμε και τις επικίνδυνες ουσίες θα δούμε ποια που οφείλονται τα προβλήματα των εργαζομένων. Όπως λέμε χρειάζονται περισσότερες έρευνες. Δεύτερη ομάδα, κίνδυνοι που κατά κύριο λόγο σχετίζονται με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, δηλαδή ανασφάλεια της εργασίας. Ξαναδιαβάζοντας την έκθεση, ξέρετε έχουμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει αυτούς τους κινδύνους πιο ορατούς. Η ανασφάλεια λοιπόν αν και στην έκθεση έχουμε γράψει πως τα παλιά κράτη-μέλη δεν είναι τόσο νέος αυτός ο κίνδυνος ε, τώρα ποια είναι η εντατικοποίηση της εργασίας περισσότερα καθήκοντα που υπομίζονται λιγότεροι άνθρωποι και υψηλότερες απαιτήσει στη δουλειά και πάλι λόγω της κρίσης λιγότεροι ε, εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τα ίδια καθήκοντα και είναι φανερό αυτό. Τέλος, βία και παρενόχληση στη δουλειά, εντάξει, αυτό είναι κάτι που ισχύει σαφώς ε, στο δημόσιο τομέα. Να σκεφτούμε τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκεί πέρα υπάρχει κίνδυνος βίας. Και τέλος, ισορροπία ζωής και δουλειάς, όπως σας είπα, το όριο ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και την εργασιακή ζωή πλέον. Χάνεται λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, ο υπολογιστής υπάρχει παντού και δυσκολεύονται να τα συμβιβάσουν αυτά τα δύο εργαζόμενοι. Μετά πιο συγκεκριμένη κίνδυνη. Τα νανοσωματίδια που έχουν αναφέρει και άλλες εκθέσεις και η Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση το έχουμε πει και στην έκθεσή μας διαταρακτές διαταράκτες μας συγχωρείτε ενδοκρινολογική ενδοκρινική και υπάρχουν κάποιες ενεργήσεις για να καταπολεμηθεί αυτό αλλεργίες κίνδυνοι που σχετίζονται με παγκόσμιες επιδημίες και εδώ πέρα έχουμε ένα μείγμα παραδοσιακών ε, εργασιακών κινδύνων με κινδύνους δημόσιας υγείας. Στην παράγραφο τη σχετική περιγράφουμε διάφορες κρίσιμες υποδομές μπορούν να κινδυνεύσουν εάν έχουμε μια παγκόσμια επιδημία και πολλοί εργαζόμενοι π.χ. από τις υπηρεσίες ε, ε, διάσωσης μπορεί να αντιμετωπίζουν τέτοιους κινδύνους. Επίσης, ηλεκτρομαγνητικά πεδία και η σχετική κίνδυνη. Αυτό σχετίζεται και με το ότι οι άνθρωποι πλέον γνωρίζουν περισσότερο τους κινδύνους. Τους πιθανούς κινδύνους π.χ. σκεφτείτε των κινητών, που κατά οποίο ακόμα είναι υποσυζήτηση. αλλά καθώς έρχονται οι έρευνες μάλλον θα έχουμε επίπτωση στην υγεία των χρηστών ε, όταν έχουμε μακροχρόνια έκθεση. Τέλος, αϊφόρες πηγές ενέργειας, δηλαδή η παραγωγή ενέργειας γίνεται όλο και πιο αποκεντρωμένη και οι κίνδυνοι, όταν μιλάμε για κινδύνους, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποιοι πολίτες θα κινδυνεύουν όταν η ενέργεια παράγεται πιο αποκεντρωμένα. Επίσης, γίνεται πιο ε, συγκεκριμένες ομάδες τώρα κινδύνου. Ε, έχουμε τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους. Μετά έχουμε αυτούς που είναι στο κατώτερα στρώματα, θα λέγαμε, της αγοράς εργασίας μετανάστες, παράνομοι, επισφαλείς εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι. Ε, βλέπετε πως όλο και περισσότερο ξεκινάνε αυτοαπασχολούμενοι νέοι άνθρωποι. Συνήθως, ε, καμιά φορά αφού απολυθούν, μια αναλλακτική λύση είναι να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Αλλά να σκεφτούμε τους κινδύνους, πραγματικά η ομάδα αυτή κινδυνεύει. Και βεβαίω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάλι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δύσκολα συμμορφώνονται με όλες αυτές τις απαιτήσεις. έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν από το να ασχολούνται με, την, ε, με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Επίσης θα βρείτε στον πίνακα αυτό μια σύνοψη. Έχουμε τους 12 τομείς ε, κινδύνου και προσπαθούμε να κάνουμε μια ιεράρχηση, κάτι το οποίο είναι δύσκολο βασίστε σε μια ποσοτική ε, προσέγγιση, μια συζήτηση δηλαδή ειδικών, ποιοι κίνδυνοι θεωρούμε ότι θα είναι σημαντικότεροι σε σχέση με τους άλλους. Βλέπετε στους τίτλους των στυλών έχουμε τον αριθμό εργαζομένων που εκτίθενται όταν ο αριθμός είναι υψηλός σαφώς είναι πιο σημαντικό το να δώσουμε προσοχή σε αυτό το κίνδυνο η διάρκεια της έκθεσης, αν μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου ή αν μιλάμε για 24 ώρες ή για όλο το 8ωρο. Το αποτέλεσμα, εάν η επίδραση μεγάλη ή μπορεί να οδηγεί στο θάνατο του εργαζόμενου, που είναι μάλλον μεγάλη επίδραση. Και τέλος η πιθανότητα. Εάν είναι υψηλή ή χαμηλή. Εάν τα συνδυάσουμε αυτά, βλέπετε έχουμε βάλει μια βαθμολογία μετά, που είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών, και έχουμε κάνει μια κατάταξη αυτών των κινδύνων. Εάν δείτε τη δεξιά στήλη λοιπόν, έχουμε ψηλότερη βαθμολογία την ε, σωματική αδράνεια, σκεφτείτε αυτό το οποίο σας είπα για την παχυσαρκία, τρόπο ζωής, καθιστική εργασία αυτό επηρεάζει τεράστιο αριθμό εργαζομένων. Επίσης, πολλαπλή κινδύνη, πολλαπλή παράγοντες κινδύνου, ε, αυτό που σας ενέφερα, ψυχοκοινωνικά, Και αυτό πάλι, ο συνδυασμός δηλαδή πάλι επηρεάζει πολλούς εργαζόμενους και δεν ξέρουμε ακόμα πολλά πράγματα για την επίδραση των πολλαπλών παραγόντων κινδύνου αλλά ε, του έχουμε δώσει αρκετά υψηλή βαθμολογία. αλλά τα έχουμε κατατάξει πιο χαμηλά, π.χ. οι ενέργειας, γιατί εντάξει ο αριθμός των εργαζομένων επίσης θα είναι μικρός. Βλέπετε είναι και μικρός ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται. Μετά έχουμε παγκόσμιες επιδημίες κτλ. Εντάξει. Αυτό είναι μικρό, αλλά εάν εκτεθεί ένας εργαζόμενος, είναι πιθανό πως θα είναι σοβαρό το αποτέλεσμα. έως μοιραίο. The, the, crisis, as I... Uh, λοιπόν, σκεφτόμενοι της ε, κρίσης, ε, όπως σας είπα, κάποιοι, την κρίση που διατρέχουμε ειδικά τώρα κάποιοι κίνδυνοι θα εμφανιστούν πιο έντονα. Σαφώς η ανασφάλεια της εργασίας αυτή τη στιγμή για μεγάλες ομάδες ε, σε συνδυασμό βεβαίως με την εντατικοποίηση της δουλειά και τη βία και την ε, παρενόχληση η ανασφάλεια θα αφορά κυρίως αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όχι τόσο στο δημόσιο τομέα. Η εντατικοποίηση επίσης της δουλειά, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα λόγω των σχεδίων, πρωτοβουλειών, ε, όλων αυτών των ανέργων που θα έρχονται και θα ζητάνε επιδόματα θα οδηγήσει σε εντατικοποίηση και στο, της δουλειάς και στο δημόσιο τομέα. Αυτό είναι ο πίνακας όπως σας είπα με βάση τη νέα κατάσταση. Επόμενη παρακαλώ διαφάνεια. Τελευταίος πίνακας λοιπόν στην έκθεση έχουμε συνδυάσει αυτούς τους κινδύνους με τις συγκεκριμένες ομάδες στόχους που βρήκαμε. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε να τον δείτε αυτό το πίνακα είναι από τα τελευταία κεφάλαια της ε, έκθεσης. Επιπλέον, παράρτημα στην έκθεσή μας είναι ένας πίνακας με τους 12 αυτούς κινδύνους και τα πιθανά μέτρα. Και αυτό είναι διαφορετικό. οι επιλογές από πλευράς ασκήσεως πολιτικής. Το περιγράφουμε αυτό στην σύνοψή μας. Στα, πιο... στα τελευταία κεφάλαια μπαίνουμε σε λεπτομέρειες για το τι είναι πιθανό και δίνουμε παραδείγματα ορθών πρακτικών από κάποια κράτη-μέλη. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να μιλήσουμε για ευρύτερες πολιτικές για να επηρεάσουμε το πώ θα εμφανιστούν αυτοί οι νέοι κίνδυνοι Και για το εάν δίνεται προσοχή σε νέους κινδύνους σε αυτές τις πολιτικές. Επίσης, ε, νέα νομοθεσία. Αν και ήδη ο τομέας αυτός ε, ρυθμίζεται σε υψηλό βαθμό και όπως λέμε στην έκθεσή μας μπορούμε να δώσουμε βάρος στην καλύτερη εφαρμογή της ε, υπάρχουσας νομοθεσίας. Οικονομικά κίνητρα σαφώς δίνουμε παραδείγματα. Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για κινδύνους που θα εμφανιστούν, χρειάζεται να εξελίξουμε νέα μέσα για τις ομάδες αυτές, για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες Επίσης ε, το να ενσωματωθούν αυτοί οι κίνδυνοι στην διαχείριση των ε, κινδύνων ε, υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα της εργασίας είτε με κάποιο έλεγχο των συστημάτων. καθώς βεβαίως πρέπει να έχουμε κατά νου πως πάντα βασιζόμαστε στην εμπειρία του παρελθόντος και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που θα προκύψουν και πρέπει να δώσουμε ειδικό βάρος σε αυτό. Και τέλος ε, γίνεται και η σύνθεση με την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή μπορεί να συνδυαστεί με τους κινδύνους αυτούς θα προκύψουν. Αυτή νομίζω ήταν η τελευταία διαφάνεια. Πράγματι, η τελευταία ήταν. Εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις, παρακαλώ είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ιδιαίτερως περιεκτική παρουσίαση. Ε, έχετε παρατηρήσεις. Ο κύριος Κρέμερς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά η παρουσίαση είναι, ήταν ενδιαφέρουσα και σίγουρα στηρίζεται σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη, αλλά βεβαίως ε, δίνει το έναυσμα σε ορισμένε ερωτήσει, σε ορισμένα ερωτήματα. Η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται εδώ σαν ένας μεγάλος παράγοντας κινδύνου και διαρωτώ με τι κρύβεται από πίσω. Και ως ε, ε, αιτιολόγηση δεν με έπεισε γνωρίζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση, η επιπτώση της παγκοσμιοποίησης είναι ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη εξωτερήκευση στην ε, παραγωγή, όλα ανατίθενται σε τρίτους, δίδονται υπεργολαβίες και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας συντονισμός σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής δηλαδή από το εργοστάσιο μέχρι το τέλος της αλυσίδας, μέχρι τα, τον κάδο απορριμμάτων. Πρόκειται εδώ για τον ε, συντονισμό ε, της ασφάλειας και της υγιεινής και εδώ δεν θεωρώ ότι υπόθηκαν πολλά πράγματα. Θα ήθελα να συμπληρώσετε εδώ κάτι. Και ένα άλλο σημείο. Η ασφαλής χρήση ε, συνεργάται επίσης με οι ασφαλείς οδηγίες μάλλον για προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορους εργαζόμενους ή από το τελικό καταναλωτή. Νομίζω και εδώ θα μπορούσε κανείς να πει περισσότερα πράγματα. Πριν από μερικούς μήνες παρακάλεσα την Επιτροπή να μας παρουσιάσει κάποιους αριθμούς για τα άτομα τα οποία βρίσκονται, δουλεύουν κάτω από άτυπες συνθήκες, μη χαρακτηριστικές συνθήκες. Γιατί σε ορισμένους ε, κλάδους υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι καινούργοι στο χώρο εργασίας και αυτοί ε, είναι ε, εκτεθμένοι σε πολλούς κινδύνους. Και αυτό αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε κανείς να αναλύσει περαιτέρω. Αυτές είναι οι σύντομες παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Γενικού χαρακτήρα. Εγώ, συνήθως, μιλώντας για την ανάπτυξη στο δικό μας κομμάτι του κόσμου, λέω ότι η σημερινή κατάσταση, όπως είπε και ο κύριος Κρέμερ, υπάρχουν ε, μετατοπίσεις των δραστηριοτήτων και παλιότερα είχαμε πολύ σοβαρότερα ατυχήματα, παραδείγματος χάρη ε, σε ένα εργοστάσιο καουτσούκ δούλευε ένας φίλος μου και όταν τελείωσε, όταν έφυγε τελικά, είχε ε, υποστεί πάρα πολλές ε, ζημιές στη σωματική του υγεία. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής. Και πώς, ε, είναι, τίθεται και το θέμα πώς ακριβώς ο εργαζόμενος μπορεί να επηρεάσει την κατάστασή του. Τι δυνατότητες έχει το άτομο να επηρεάσει την κατάστασή του στην εργασία. Πώς μπορεί να την επηρεάσει ε, με θετικό τρόπο. Υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση και εξαρτώνται πλέον από τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκ των άνω και επηρεάζουν την ε, κατάστασή τους στην, ε, την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας. Τι έχετε να πείτε εσείς για αυτό το θέμα. Η πρώτη ερώτηση ήταν ο συντονισμός της αλυσίδας της αλυσίδας παραγωγής ε. υπάρχει ένα συναφέ ζήτημα μέσα στην έκθεση το θίγουμε ε, με περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι στην παρουσίαση που κάναμε δίνουμε και παραδείγματα σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν και καταστάσεις ε, όπου αυξάνεται η αυτονομία των εργαζομένων και έτσι βελτιώνεται η κατάσταση ή τονώνεται ο κοινωνικός διάλογος. Επίσης το θέμα της διακυβέρνησης για την υγεία στο χώρο εργασίας, η τόνωση του κοινωνικού διαλόγου για τα κλαδικά προβλήματα. Ίσως σας βοηθήσουν τα παραδείγματα ε, σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και βλέπουμε και τις ε, συστάσεις που είναι υψηλού επίπεδου, λίγο υψηλού επίπεδου φυσικά. Τόνωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ε, παραδείγματος χάρη, τέτοιου είδους λύσεις. Ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση. Θέλεις να προσθέσεις κάτι για αυτό το θέμα. Ehm, eh, ε, ναι, σε σχέση με αυτό που μας είπε ο κύριος Κρέμερς ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι για τον συντονισμό της ε, αλυσίδας ε, δίκιο έχει, της αλυσίδας παραγωγής δίκιο έχει το λέμε μέσα στην έκθεση, κυρίως θα μιλάμε για καταστάσεις όπου υπάρχουν πολλοί αυτοαπασχολούμενοι. όπως σε πολλές επιχειρήσεις, ε, όπου η εργολάβοι ας πούμε, ε, που είναι κίνητα αφεντικά. Και στα εργοτάξια έρχονται διάφορα και παρέχουν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Εκεί είναι εκδηλά τα προβλήματα. Αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό μόνο τον τομέα το πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις θέλουν να υπάρχει καλή σχέση κόστους-οφέλους. Επειδή, δηλαδή, πρόκειται για περίπλοκα πρότυπα. Έχουμε και μετανάστες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που ε, έρχονται να εργαστούν στη Δυτική Ευρώπη. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα σε κάποιους τομείς. Εσείς μιλήσατε για τα, το καουτσούκ. Ναι, είναι πολύ υπαχθής η εργασία. Και έρχονται κάποιοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ουκρανία παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολύ ε, περίπλοκη η κατάσταση και ο συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες ε, μικρές επιχειρήσεις ε, δημιουργεί εξίσου μεγάλο πρόβλημα. Ακόμη και για τους ίδιους εργαζομένους. Um, Υπήρχε και ένα τελευταίο ερώτημα για τους εργαζόμενους, τι μπορούν εκείνοι να κάνουν για να βελτιώσουν την κατάσταση. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα παραδείγματα και στην ίδια την έκθεση και στα παραρτήματα όπου απομονώνουμε κάποιους τομείς συνάδελφος μπορεί να σας δώσει παραδείγματα. Στην αστυνομία παραδείγματος χάρη προσπαθούν να ε, ρυθμίσουν το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης ε, έρχονται σε επαφή με τον ε, εργοδότη ή με τον προϊστάμενο Ε, τέλος πάντων ε, νομίζω ότι έρχονται άμεσα, δηλαδή σε επαφή εργαζόμενοι με τον προϊστάμενο ή με τον εργοδότη και τα λύνουν μόνο τους τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ε, μπορείτε να εμβαθύνετε τη μελέτη όσοι θέλετε. Ε, σας ευχαριστούμε. Α, α, η Επιτροπή θέλει να μας πει κάτι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρετε, ήρθα από το Λουξέμβουργο και δεν ήρθα μόνο για να ακούσω τη μελέτη, θέλω να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχά, ε, να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία ε, για να διεξαχθεί αυτή η μελέτη. Τώρα, για τους αναδυόμενους κινδύνους, ε, δηλαδή το ίδιο το αντικείμενο της έκθεσης, θα πρέπει να σε ενημερώσουμε κι εμείς τι κάνουμε στη δική μας υπηρεσία για να ξέρετε πώς ε, αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα των αναδειωμένων κινδύνων. Πρώτον, υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν λειτουργικές δομές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Ε, τεχνικές επιστημονικές ομάδες εργασίες ε, στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την ομάδα εργασίας για τις χημικές ουσίες. Να, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μεταξύ άλλων. Επιστημονική Επιτροπή για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης ε, για την αξιολόγηση των χημικών ουσιών επικινδύνων υλικών αλλεργιογόνων, διαταρακτών του συστήματος, του ενδοκρινικού συστήματο κτλ και ε, ε, ε, η ενιαία υπηρεσία για την επιθεώρηση εργασίας. Έχουμε και στον Πιλμπάτ σχετική υπηρεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και η δική τους εντολή είναι η συλλογή των δεδομένων και κοινοποίησή τους. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια ζητήματα τη έκθεση. Νανοτεχνολογία. Η γάμα δέλτα μου ε, εκπροσωπεί την ομάδα της για τις Νανοτεχνολογίες. Ε, υπάρχει ομάδα αναθεώρησης ε, διυπηρεσιακή για το περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Παρακολουθούμε από κοντά τις εργασίες αυτών των ομάδων για τα ψυχολογικά ζητήματα, ψυχοκοινωνικά ζητήματα. Δεν είμαι και τόσο ειδικό, αλλά τέλος πάντων. συνδέονται με τα ε, θέματα ψυχικής υγείας ε, γενικότερα ε, από τη γάμα δέλτα καταναλωτών που έχει τη βασική ευθύνη έγινε στις 13 Ιουνίου πέρσι και σχετική διάσκεψη και μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν να διοργανωθούν θεματικά σεμινάρια μεταξύ των οποίων και ένα για αυτό το θέμα στην αγορά εργασίας δηλαδή και τους κινδυνούς ε, για την ε, ψυχική υγεία. Κάποια στιγμή το 2010 θα γίνει αυτό. Ξέρετε, τώρα έχουμε και αυτή την διαδικασία ε, ε διαγωνισμών για την συλλογή πληροφοριών. Δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε τη διαδικασία. Ένα παράδειγμα για την οδηγία, για την εφαρμογή της οδηγίας ε, για τις ε, χημικές ουσίες και τις κατοικινογόνες ουσίες. Θα εξετάσουμε και το θέμα της αντικατάστασης κάποιων χημικών ουσιών ο τίτλος έκθεσης είναι «Ποια είναι η επίπτωση στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία με την αυξανόμενη χρήση ε, των υπολογιστών και γενικά των εργαλείων πληροφορικής». Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που ε, τονίζονται μέσα στην έκθεση. Ε, επίσης, οι επιθεωρητές εργασίας, για τους επιθεωρητές εργασίας, το 2009 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός υπηρεσίε των επιθεωρητών εργασία ασχολούνται με αυτό το θέμα της υγείας και της ασφάλεια ε, στην εργασία ε, και ε, κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας θα διοργανωθεί διάσκεψη για τους ψυχοκοινωνικού κινδύνους στο χώρο εργασίας. Τον Ιούλιο του 2009 θα γίνει διάσκεψη στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της ΓΔ Απασχόληση. Θα συμμετάσχουν φυσικά και άλλες υπηρεσίες επιτροπής αλλά το θέμα θα είναι το στρες στο χώρο εργασίας. Αυτή... Κλείνοντας να πω ότι καλωσορίζουμε αυτήν την έκθεση. Είναι πολύ καλό εργαλείο για να διευρύνουμε τη βάση πληροφοριών που έχουμε και που χρειαζόμαστε για να λάβουμε αποφάσεις. Ποιες είναι οι λογικές εναλλακτικές ε, λύσεις για την πολιτική που θα ακολουθήσουμε, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, χρειαζόμαστε χρόνο για να αποφανθούμε ότι να, αυτός είναι ένας συγκεκριμένος αναδυόμενος κίνδυνος, όπως με τις νέες τεχνολογίες που σας έλεγα. Ένα παράδειγμα είναι αυτή η μελέτη που σας είπα για την ε, χρήση των ε, εργαλείων ε, πληροφορικής για τις τηλεπικοινωνίες και των υπολογιστών. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά πριν από αυτό Πρέπει να γίνει διαβούλευση με ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων, για να, αλλιώς δεν μπορούμε να λάβουμε μια σωστή απόφαση. Σας ευχαριστούμε. Πέρα στη συζήτηση και θα μας ξαναπασχολήσει το θέμα. Χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μελέτη για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Δεν έχουμε άλλα σημεία στην μερίσια διάταξη. Να σας ανακοινώσω απλά ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 2 Μαρτίου, στις 3. Δευτέρα είναι. Και μέσα στη βδομάδα θα μας επισκεφθούν και οι εκπρόσωποι της μελλοντική Σουηδικής Προεδρίας. Οι συντονιστές ε, να παραμείνουν, ε, γιατί θα κάνουμε τη συνεδρία των συντονιστών τώρα. Ευχαριστώ.